Dear colleagues. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σα ημέρα. Και πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου, τα βαθύτατα συλληπιτήριά μας για τα θέματα των ε, αποτρόπαιων επιθέσεων στο Παρίσι. Υπενθυμίζω δε σε όλους τους συναδέλφους ότι στις 3 το μεσημέρι προβλέπεται μια έκτακτη σύνοδος, σύντομη σύνοδος στην Ολομέλεια για να αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας και να εκδηλώσουμε την αλληλική μας με το γαλλικό και τις γαλλικές αρχές. Και προχωρώ στην ημερήσια διάταξη. Για να ρωτήσω εάν εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Πρόκειται για μια δημόσια κρόση για την ε, πιθανότητα παράτασης των ε, θητιών των επικεφαλής των επικοπτικών αρχών, όπως ξέρετε. αποφασίστηκε το Σεπτέμβριο η παράταση της ε, θητείας των προέδρων, των απερχομένων προέδρων της τρεις ε, εποπτικές αρχές και χρειάζεται η επικύρωση αυτής της απόφασης για τριετή παράταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλέπετε λοιπόν την 1η Δωδεκάτου να γίνει σχετική ψηφοφορία στην Επιτροπή μας μετά τις ακροάσεις και στην Σύνοδο του Στρασβούργου στη συνέχεια θα επικυρωθεί και από την Ορλομέλεια. Επίσης παρατείνεται για τρία χρόνια και η θητεία των εκτελεστικών διευθυντών της ΕΤΑ και της ΕΣΜΑ και βεβαίως θέλουμε να συζητήσουμε τα επιτεύγματα και τα καθήκοντα των αρχών για δε την ε, ΙΟΠΑΣ, για την ε, υπηρεσία ε, ασφαλίσεων και συνταξιοδότησης χρειάζεται κύρωση από το Κοινοβούλιο του διορισμού του νέου διευθύντη και στην διαδικασία αυτή αναλαμβάνει δράση η ΕΚΟΝ. Σήμερα λοιπόν διεξάγονται οι ακροάσεις με τους απερχόμενους ε, επικεφαλής που πρόκειται να, των οποίων πρόκειται να παραταθούν οι θητείες. Βλέπουμε με χαρά τον κύριο Άντρεα Ερία εδώ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και θα ήθελα να του δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Μετά θα αρχίσουν οι ερωταπαντήσεις. Αλλά πριν αρχίσω θα ήθελα, να αρχίσετε θα ήθελα να σας συγχαρώ για το έργο που έχει επιτελέσει η ΕΤΑ στο διάστημα αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν επίσης πάρα πολύ καλή η συνεργασία σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο. Thank you ε, Ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτο. Σας ευχαριστώ όλους ε, για, που με έχετε ενώπιον σας στην αρχική μου δήλωση στην Επιτροπή σας κατά την ακρόαση επιβεβαίωσης επικύρωσης πριν από πέντε χρόνια είχα πει ότι θα κάνω την μπορώ για να γίνουν οι αλλαγές που είχε ζητήσει ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα για να ανταποκριθούμε στην ε, χρηματοπιστωτική κρίση και ότι θα υπάρξει αποφασιστική δράση για να ενισχύσουμε τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα να υπάρξει ένα πραγματικό ενιαίο εγχειρίδιο για να υπάρξουν οι μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα και να αναπτύξουμε τα νέα εργαλεία για να υπάρξει πραγματική σύγκληση στις εποπτικές πρακτικές και νέα προσοχή σε θέματα καταναλωτών. Δεν μπορώ να πω σήμερα ότι τα έχουμε επιτύχει όλα, αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή του Τραπεζικού Τομέα, η EBA, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες έχουν ενισχύσει την κεφαλιακή, την θέση, που τώρα είναι ισχυρότερη από τις αντίστοιχες των ΗΠΑ. Επίσης έχουμε ουσιώδη, έχουμε επιτύχει ουσιώδη γνωστοποίηση των στοιχείων για τις τράπεζες, κάτι που θα ε, συμβάλλει στο να υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό τομέα και την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιεύσουμε την ε, προσπάθεια διαφάνειάς μας. Θα γνωστοποιήσουμε πάνω από 13.500 στοιχεία δεδομένων για κάθε τράπεζα, για περισσότερες από 100 τράπεζες. Το ενιαίο εγχειρίδιο αφορά βασικούς τομείς της επιτήρησης και της εξυγίανσης. Έχουμε πολλές κατευθύνες γραμμές και ερωτήσεις τις οποίες καταφέραμε να ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Και επίσης έχουμε ε, ε, ξεκινήσει και διαδικασίες για παράβαση του νόμου καθώς και διαιτησίες για να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά. Παρά το ότι ξεκινήσαμε αργά τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε σημειώσει ισιώδεις προόδου για θέματα καταναλωτών έχουμε αντιμετωπίσει θέματα που προκύπτουν από καινοτόμα προϊόντα και έχουμε και δικέ μα κατευθυντήριε γραμμέ, ιδιαίτερα για την υπόθηκα δάνεια και για την διακυβέρνηση και εποπτεία των ε, ε, προϊόντων. Βεβαίω πρέπει να αλλάξουμε εστίαση ούτω ώστε να έχουμε πιο εκλεπτισμένη ε, προσοχή στην ενιαία αγορά των 28, για να, των 28 ε, κρατών για να συνδέσουμε ε, τα κράτη εντός και εκτός της Ευρωζώνης. αν επιβεβαιώσετε την αποστολή μου θα αναλάβω την εξή δράση. Πρώτον, θα αναπτύξουμε μια, ένα θεματολόγιο για να υπάρξει σύγκληση στις πρακτικές επιτήρησης και εξυγίανση. Άρα θα χρειαστούμε νέα εργαλεία. Για παράδειγμα να ελέγχουμε και τα αποτελέσματα όπως κάνουμε τώρα στη δουλειά μας για την σταθερότητα και αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού με στάθμιση κινδύνου και την αναθεώρηση ορισμένων παλιών εργαλείων όπως τα τεστ αντοχής και η κατάρτιση των ελεγκτών και περισσότερος εστιασμός, περισσότερη εστίαση σε θέματα που έχουν να κάνουν με τους κυβερνοκινδύνους. Επιπλέον πρέπει να δούμε πώς επηρεάζονται από τη δράση της ε, ρυθμιστικής αρχής οι, οι αγορές στον τραπεζικό τομέα. Γενικά, οι μελέτες αντικτύπου εξέτασαν ε, πώς λειτουργούν τώρα οι τράπεζες και την δομή των ισολογισμών. Αλλά αυτά πρέπει να αλλάξουν μετά τις ε, αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Άρα πρέπει να καταλάβουμε Εάν αυτέ οι αλλαγέ που προκαλούν οι νέοι κανόνε προκαλούν παρενέργειε και αν οι προσπάθειε του κλάδου για να ελαχιστοποιηθεί το ρυθμιστικό βάρο δημιουργούν νέου κινδύνου στον τραπεζικό ή προκαλούν μετατόπιση σε άλλα τμήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό είναι ουσιώδε για να διατηρήσουμε τι τεχνικέ προδιαγραφέ και κατευθυντήριε γραμμέ. Αλλά όταν χρειάζονται αλλαγέ, θα προσπαθήσουμε να δούμε και τα στοιχεία που πρέπει να μας οδηγήσουν να αλλάξουμε την πρωτογενή νομοθεσία και να δούμε και αν υπάρχουν ακαμψίες ορισμένα σημεία. Επίσης οι αναλύσεις μας πιστεύουμε ότι πρέπει να ασχοληθούν με την πολυπλοκότητα του νέου ρυθμιστικού πλαισίου και την σωστή εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας. Ο τρίτος τομέας είναι να ασχοληθούμε περισσότερο με την προστασία των καναλωτών, ιδιαίτερα στα πλαίσια τη ε, χρηματοπιστωτική καινοτομία. Η ψηφιακή τραπεζική δραστηριότητα θα είναι μια πρόκληση για του επιτηρητέ, για του επόπτε, του επόμενου τομεί. Δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικοί και να εμποδίσουμε την χρηματοπιστωτική καινοτομία, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τελικοί χρήστε ε, προστατεύονται επαρκώ. Και ο κύριο τομέα θα είναι οι υπηρεσίες πληρωμών. Και ε, χαιρετίζουμε τι εντολέ που προκύπτουν από το PSD2 την οδηγία PSD του, αλλά και υπάρχουν και άλλοι τομεί εργασία, όπω για παράδειγμα ο δανεισμό μεταξύ ομοτήμων που πρέπει να μα απασχολήσει. Τώρα, επειδή δεν έχουμε επαρκή προπολογισμό, δεν είμαστε σε θέση να ε, αναπτύξουμε τι δραστηριότητέ μα όπω θα θέλαμε. Για παράδειγμα, οι προσπάθειέ μα να έχουμε ένα φιλόδοξο ε, σχέδιο κατάρτισης των επιτηρητών. Όλα αυτά εμποδίζονται από τους περιορισμούς που έχουμε. Η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα προϋπολογισμού ε, μας ε, ε, ενθαρρύνει πολύ, αλλά τα προβλήματα παραμένουν, θα χρειαστεί περισσότερη δράση, πιο ριζική δράση. Πιστεύω ότι κατά την πρώτη μου θητεία ως ε, Προέδρου δημιουργήσαμε ένα κλίμα καλού διαλόγου με τα τρία θεσμικά όργανα. Αυτό γίνεται σε διάφορα επίπεδα, τεχνικός άτυπος διάλογος, πρόορη προειδοποίηση για ευαίσθητα θέματα, συμμετοχή σε διάφορες κοινέ εκδηλώσεις και επίσημες ακροάσεις. Ως επικεφαλής μια αρχή ε, που δίνει μεγάλο βάρος στην ανεξαρτησία της, πιστεύω στην διαφάνεια και τη λογοδοσία και ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτή την καρποφόρα σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Ένα λεπτό αναερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση. Ο κύριος Μπάλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έφυγε και το πρώτο μισό μου λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και καλώς ήρθατε κύριε Ανδρία. Πολύ σύντομα έχω δύο ερωτήσεις. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον θα μπορούσατε παρακαλώ να μας εξηγήσετε πώς βλέπετε προσωπικά την συνεργασία στον χώρο της τραπεζικής εποπτείας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχετε μια πρώτη εμπειρία από τη δουλειά ενός περίπου έτους. Χρειάζεται όμως περισσότερη σαφήνεια. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Και δεύτερη. Ναι, και κάνατε λόγο για την πολύ καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ και εγώ ότι είναι καλή, αλλά υπάρχουν ε, κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι λένε ότι συνεργάζεστε πολύ στενά ιδιαίτερος με το Συμβούλιο. Τι θα πείτε σε αυτές τις επικρίσεις, τι θα απαντήσετε. Τι κάνουν δηλαδή οι εποπτικές αρχές, είναι πολύ πιο στενή συνεργασία τους με το Συμβούλιο προς την εποπτεία των τραπεζών και την εποπτική λειτουργία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάλτς για την ερώτηση. Όντως είναι κρίσιμη η πρώτη ερώτηση στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού. Ε, φυσικά θα ήθελα να σημειώσω έχουμε πολύ καλέ σχέσει σε κάθε επίπεδο επαγγελματικό και εργασίας. Η πεποίθησή μου είναι, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από τις πρώτες ε, εμπειρίες από τον αποπτικό μηχανισμό, ότι ε, θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και δεν μπορούμε βεβαίω να έχουμε μια εποπτική αρχή η οποία θα εφαρμόζει σε διαφορετικές τράπεζες διαφορετικούς κανόνες ανάλογα με τη δικαιοδοσία. Θα πρέπει να προχωρήσουμε προς περισσότερη εναρμόνιση. Άλλωστε αυτό το είδαμε και στην συζήτηση που έγινε για τις ε, ιδιαιτερότητες τις εθνικές και όλα αυτά θα μας οδηγήσουν σε μια πολύ πιο ουσιαστική εναρμόνιση. Με τρεις επιλογές, τρεις εναλλακτικές. Για μένα ε, η καλύτερη εναλλακτική θα ήταν ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για όλη την ενιαία αγορά, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα διαφυλασσόταν και η ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς τη ενιαία αγορά. Δεύτερον, αυτό που αρχικά είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη θέσπιση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, να έχει δηλαδή ρυθμιστικέ αρμοδιότητε ο ίδιο ο μηχανισμό. Αυτό θα επέλυε βέβαια τις δυσκολίες, τα προβλήματα στην νευροζώνη, αλλά θα οδηγούσε σε ένα εγχειρίδιο κανόνων δύο ταχυτήτων. Και θα παγίωνε με τον τρόπο αυτό και τα διαφορετικά κλιμάκια μέσα στην εσωτερική αγορά, τις διαφορετικές κλίμακες πρόοδου. Πράγμα αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο. Και η τρίτη, που θα είναι η μόνη λύση που θα μας μείνει αν δεν ευρεθούν ε, λύσεις σε θεσμικό επίπεδο, να οδηγηθούμε σε λιγότερο διαφανή εργαλεία ε, εγχειρίδια εποπτεία, εσωτερικέ κατευθυντήριε γραμμέ που πολλέ φορέ δεν έχουν καμία διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται εμεί να πιέσουμε από πλευρά μα για ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η επισήμανσή μου σχετική με συγκλίνουσα εποπτική πρακτική έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι οι τράπεζε βρίσκονται υπό την εποπτεία τη ΕΚΤ πολλές φορές έχουν δραστηριότητες και εκτός της Ευρωζώνης και άρα αυτός ο ρόλος της γέφυρας μεταξύ του ενιαίου αποπτικού μηχανισμού και της έξω ζώνης, της έξω περιοχής, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για την άλλη σας παρατήρηση δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Στο σχόλιο. Δεν θα συμφωνήσω στο σχόλιο ότι συνεργαζόμαστε καλύτερα με το Συμβούλιο από ότι με το Κοινοβούλιο. Εγώ προσωπικώς πιο πολύ χαίρομαι τις συζητήσεις με το Κοινοβούλιο. Γιατί στο Συμβούλιο σε ένα βαθμό αντικατοπτρίζονται οι εθνικέ θέσει, που τόσοι άλλω βλέπω και στο τραπέζι του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο πολύ μου αρέσει η ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο. Ωστόσο υπάρχουν πολλές δίωδοι ανταλλαγής, πληροφοριών, διαλόγου και έχουμε νομίζω και συμφωνήσει με τους αδέρφους και, με τη, και τη ΣΕΣΜΑ και τη ΕΙΟΠΑ να προχωρήσουμε αναζητώντας διαφορετικές αναλλακτικές και σε άτυπες ανταλλαγές απόψεων αλλά και σε ενημέρωση άτυπη με υπομνήματα που θα μπορούσαμε να σας αποστέλουμε για να ενημερώνεστε και βέβαια θα θέλαμε και εμείς να βλέπουμε τις δικές σας θέσεις και απαντήσεις στις προτάσεις μας. Σας ευχαριστούμε ο Πέτρος Ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση σχετίζεται σε αυτό που είπατε στην εισαγωγική σας ε, ομιλία ε, διαφοροποίηση των εποπτικών αρχών. Εδώ είναι δημόσια συνεδρίαση. Θέλω να γραφτεί και στα πρακτικά ότι η ΕΜΠΑ θεωρεί ότι δεν μπορεί να αναπτύξει την εποπτική του δραστηριότητα όπως θα ήθελε διότι δεν έχει επαρκή προϋπολογισμό. Πρέπει να το τονίσουμε. Ίσως να το καταλάβει και εκείνη η γνώμη. Γιατί αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που θέλαμε. Θέλαμε οι τρεις εποπτικές αρχές όταν δημιουργήθηκαν να μην είναι μόνο στα χαρτιά εποπτικές αλλά στην πράξη. Και αν δεν υπάρχει επαρκής προπολογισμό, αν δεν υπάρχει επαρκής κατάρτιση, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο περισσότερες πιστώσει χρειάζεστε ούτως ώστε να κάνετε τα καθήκοντά σας εποπτείας και κατάρτιση του προσωπικού σας όπως τα θέλατε. Δεύτερη ερώτηση. Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την ομοθεσία για την ε, ενοποίηση των κεφαλαίων προσπαθούμε να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Ξέρουμε ότι 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρομεσαίες. Ξέρουμε ότι δημιουργούν το 67% των νέων θέσεων εργασίας. Έχουν λοιπόν έναν ειδικό ρόλο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελευταία κρίση δεν ε, προκάλεσαν την κρίση αυτές οι χρηματοδοτήσεις ούτε για το ενιαίο κεφάλαιό τους. Προσπαθήσαμε να ε, ευνοήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Άκουσα ότι διάφοροι εκπρόσωποι της ΕΜΠΑ και εσείς μόλις είπατε ότι με βάση τα στοιχεία σας σκέφτεστε ότι θα έπρεπε να μειωθεί αυτή η εύνοια προς μικρομεσαίες. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα είχε βλαβερά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Σίμων για την πρώτη σας ερώτηση. Να σας δώσω το παράδειγμα των ασκήσεων, των πρακτικών ασκήσεων. Εκεί προσπαθούμε να έχουμε ένα οργανωμένο σύστημα με ένα ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα ώστε να μπορούν όλοι οι υπεύθυνοι ανά την Ένωση να το εξετάσουν με τον ίδιο τρόπο. Με υλικό για τις πρακτικές ασκήσεις που θα χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο οι εθνικές αρχές και την πιστοποίηση αναλόγως. Οπότε κάθε επόπτης στην Ευρώπη να έχει τα ίδια εργαλεία. Και έχουμε και εταιρική σχέση με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα των Πανεπιστημίων και πολύ επιγραμμική εκπαίδευση online ώστε όλοι σε όλους τους τομείς που ενδιαφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν πρόσβαση. Βεβαίω, για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε πόρου. Και επειδή έχουμε περιορισμούς, σκεφτήκαμε κατά πόσο μπορούν και οι εθνικές αρχές να συνεισφέρουν. Διότι ο προπολογισμό που σε εθνικό επίπεδο αποδίδεται στι ε, στις πρακτικές ασκήσεις θα περάσει απλώς στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θέλουμε πρόσθετα κονδύλια Μιλάμε για ένα ποσό 2 εκατομμύρια συνολικά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να έχουμε προς τα κονδύλια, δεν μπορούμε να τα έχουμε. Ούτε θέλουμε ξεχωριστή χρηματοδότηση από τις εθνικές αρχές με δημοσιονομική γραμμή. Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια δραστηριότητα από διαφορετικό προπολογισμό πέρα από το δικό μα και δεν μπορούμε να χρεώσουμε και κάποιε αμοιβέ, απολαυέ για αυτέ τι μαθητείε. Δεν θα μπορούμε να το κάνουμε λοιπόν αν δεν γίνει έτσι και θα είναι κρίμα. Ω προ την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτή τη στιγμή κάνουμε μια μελέτη, την οποία θα φροντίσουμε να σα αποστείλουμε του χρόνου, όπω ζητήθηκε, και βασιζόμαστε σε πολύ συγκεκριμένα πρακτικά στοιχεία. Συμφωνώ μαζί σα ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν ήταν το επίκεντρο τη κρίση, δεν ήταν από τα αίτια, όμω προφανώ επηρεάστηκε η οικονομική τους κατάσταση και πολλά από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν να κάνουν με το πόσο τεθειμένες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουμε τελειώσει τη μελέτη βέβαια, αλλά μερικά ενδεικτικά στοιχεία είναι ότι για το κεφάλαιο, το δευτερογενές κεφάλαιο δεν ήταν πολύ απλό για την στήριξη των μικρομεσαίων να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, ο δεύτερο, δευτερεύον παράγοντας από τη στιγμή που άρχισε να ισχύει δεν εξυπηρέτησε την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Υπάρχουν όμως ε, χαμηλότεροι παράγοντες κινδύνου στα χαρτοφυλάκια των ε, μικρομεσαίων και ε, μικρότεροι παράγοντες συσχετισμού, λόγοι συσχετισμού βάσει του μοντέλου εσωτερικού σχεδιασμού. Πάντως, βλέποντας το ποσοστό κινδύνου που υπάρχει στην συναλλαγή, Υπάρχει ενδεχομένω υπερχρέωση στο κεφάλαιο των μικρομεσαίων ανάλογα με το χαρτοφυλάκιό τους. Αυτά είναι τα στοιχεία που λίγο πολύ θα σας παρουσιάσουμε. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Κάποιες φορές υπερβάλλουμε ως προς τον αντίκτυπο των ρυθμιστικών απαιτήσεων στην, ε, στο δανεισμό και οι παράγοντες που κρίνουν το δανεισμό είναι πιο πολύ το κατά πόσον ε, υπάρχει παράγοντας κινδύνου του αντισυμβαλωμένου και τι πίστοση ζητάει. Αυτό περισσότερο επηρεάζει το επίπεδο της ζήτησης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα πρέπει να βέρνουμε βέβαια τι θα γινόταν και αν απουσίαζαν αυτές οι συνθήκες. Η κυρία Σούνπερ. Ευχαριστώ σας ευχαριστούμε για το σχεδιασμό των κανόνων επίπεδου 2 στην περασμένη σας θητεία και σας επενώ και εσάς και του συνεργάτες σας για αυτή τη δουλειά. Αλλά στις νομοθετικές μας προτεραιότητες ε, ήδη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και άλλα εργαλεία και να ενισχύσουμε το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων με τη συμμετοχή των εθνικών αρμόδιων αρχών. Θα αρχίσουν λοιπόν να έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία τα έγγραφα που ετοιμάζεται. Τι διαφάνεια θα παράσετε στους ε, ε ενδιαφερομένους για την εφαρμογή των κανόνων και τι ε, κατεύθυνση θα μπορούσατε να δώσετε στις εθνικές αρχές, στις εθνικές αρμόδιες αρχές και όσους ενεργοποιούνται στην αγορά. Επίσης, τι μέτρα μπορείτε να λάβετε εσείς από τη θέση σας για να αποφύγετε την ε, πολιτική επιρροή που μπορεί να έχουν τα μέλη του Διοικητικού σας Συμβουλίου. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ήδη αλλάζει η προσέγγιση και βλέποντας το θεματολόγιο από εδώ και μπρος μπορώ να σας πω ότι το 2016 μας απασχολήσει ακόμη για σημαντικό κομμάτι η παραγωγή προδιαγραφών και προτύπων. Από το 2017 και μετά θα αρχίσουμε να αποδεσμεύουμε πόρους για να κινηθούμε προς την ε, ουσιαστική υλοποίηση και την σύγκληση των εποπτικών πρακτικών και εκεί θα είναι η κύρια πρόκληση για μας γιατί το σύστημα διακυβέρνησης που έχουμε περιπλέκει πολύ τη δομή και τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζονται νέα εργαλεία η συγκριτική αξιολόγηση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επί παραδείγματι στα, ο ενεργητικό το σταθμισμένο προς τον κίνδυνο, αλλά και σε άλλους τομείς. Ε, αυτό που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε φέτος ήταν μια, ήταν μια έκθεση για την εποπτική σύγκληση και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει και το κυριότερο εργαλείο με το οποίο μπορούμε, επικοινωνώντας μαζί σας, να σας δείξουμε ποια είναι τα σημεία ε, στα οποία εντοπίζουμε προβλήματα και, δίνουμε, και κάνουμε προτάσεις. Και βεβαίως μπορεί κάποια πράγματα να μην λειτουργούν καλά επειδή η πρωτογενής νομοθεσία δεν μας το επιτρέπει. Δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε προς τη σύγκληση. Θα το έχω ξαναπεί, είχαμε το θέμα της αναλογικότητας ως προς τις αμοιβέ, εκείνη τη διάταξη που ίσως μας απασχολήσει αργότερα στη συζήτηση. Αυτό είναι μια άλλη γραμμή διαλόγου δηλαδή. Όταν βλέπουμε αποκλίνουσες προσεγγίσεις από το λόγο με τον οποίο υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο ή οδηγίες, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και προσκόμματα ω προς τη σύγκληση. Για τα για τα πρότυπα, ε, βεβαίως είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Είναι στο Διοικητικό μα Συμβούλιο και ανοίγοντα μια παρένθεση θα ήθελα να πω ότι στη διακυβέρνηση, στο σύστημα τη διακυβέρνηση που έχουμε βλέπουμε κάποιε δυσκολίε και αισθανόμαστε δυσφορία και αντιλαμβάνομαι βεβαίω ότι του κανόνε τους έχει επιβάλει το Συμβούλιο άρα δεν μπορώ και να του αμφισβητώ αλλά υπάρχουν περιπτώσει όπου αποχέ που διατυπώνονται στι διαπραγματεύσει. στο δικό μα το Διοικητικό Συμβούλιο ε, και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 23 ψήφους υπέρ, 5 αποχές και καμία ψήφο κατά και άρα ε, αποτύχαμε στην εξασφάλιση απαρτίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε γιατί οι ε, κατευθύνες γραμμές τις οποίες εκείνη την ώρα δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν. Και έτσι... Φυσικά θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε ε, με σκληρή δουλειά, κάνουμε ό,τι μπορούμε και για να ε, αποφύγουμε χάρη σε ένα διάλογο με τα κράτη-μέλη εθνικές τοποθετήσεις, έτσι ώστε και το Συμβούλιο να έχει μια ισορροπημένη τοποθέτηση για να προχωρήσουμε προς την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Αλλά βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται και από τις διαδικασίες εγκρίσεως. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουλάχ. Ευχαριστώ κυρία που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί σα και ευχαριστούμε για όσα κάνατε αυτά τα χρόνια όταν αναλάβαμε την ευθύνη με κάποιου άλλου που δεν είναι πια εδώ βέβαια, αλλά όταν αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε, να ιδρύσουμε αυτέ τι αρχέ. ήταν πολύ δύσκολη απόφαση και πριν την Τραπεζική Ένωση ξέραμε τι ελλείψει υπάρχουν στη διακυβέρνηση τη αρχή ιδίω που με πολύ ε, ταλαντούχο τρόπο διευθύνεται. Κάποια πράγματα που με ανησυχούν τελευταίως, ιδίως η διασύνδεση μεταξύ των μέτρων επίπεδου 1 και όσων μπορεί να σας ζητηθούν τελικά, νομίζω. Δεν είναι μυστικό ότι το κείμενο για τη διευθυντική μεταρρύθμιση των τραπεζών υπάρχει μια παραπομπή σε μια από τις συμβαστικές λύσεις που προτείνονται, που είναι κάπως δυσβάχτης τακτή για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ίσως κάποια κράτη να απόσχουν και το κείμενο να μην μπορέσει να εφαρμοστεί. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι σκέφτεσαι για την κατανομή μεταξύ επίπεδου 1 και 2. Μπορείτε να αλλάξετε την ε, διακυβέρνηση του επίπεδου 2. Ε, πιστεύετε ότι πρέπει να σκεφτούμε άλλες ιδέες. Τι μας προτείνατε να λάβουμε υπόψη. Σε Γενικέ γραμμές, ο ασχετισμό επίπεδου 1 και 2 είναι σημαντικό ζήτημα. Προσωπικός. Πιστεύω ότι όταν η Επιτροπή διεξάγει αναθεώρηση, όπω προσχέθηκε ο Επιτροπό Χίλ, για τη μεταρρύθμιση των τραπεζών, θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Υπάρχουν τομείς όπου στο επίπεδο 1 οι κανόνες είναι υπερβολικά λεπτομερείς ίσως και είναι δύσκολο να εφαρμοστούν πρακτικά στην αγορά, στις αγορές και κάποιες, ε, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί συμφωνία στο επίπεδο 1 οπότε το δύσκολο θέμα παραπέμπεται εύκολα στο επίπεδο 2 Σίγουρα σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε σημασία, να έχουμε ένα νέο εγχειρίδιο κανόνων που να είναι και σαφές και εξισορροπημένο και με τις ε, κατάλληλες αρχές ώστε να υπάρχει και το σωστό επίπεδο λεπτομεριών στο επίπεδο 2. Πάντα δίνω και το παράδειγμα της υποβολής εκθέσεων. Νομίζω το μεγαλύτερο ζήτημα ε, της επίσημης εφημερίδας είναι τα δικά μας τα πρότυπα και αν ε, υποβάλαμε εκθέσεις χωρίς να δημοσιεύονται στην ε, επίσημη φυρίδα δεν θα είχε και νόημα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που αποσχολεί και τι τεχνικέ αρχέ και θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε κάπως Τώρα για τι διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις και το πώ πρέπει να γίνουν αυτά που αναφέρατε. Σε γενικέ γραμμέ, στηρίζοντα συμπεράσματα τη έκθεση Λίκανεν, νομίζω ότι και εξορροπημένοι είναι και διατηρεί τα γνωστά μοντέλα των τραπεζών αντιμετωπίζοντα και του ε, ανάλογου κινδύνου. Απλώ είδαμε και πολλέ εθνικέ μεταρρυθμίσει που δεν συντονίστηκαν επαρκώ ω σήμερα. Όμω οι προποθέσει υπάρχουν για να γίνουμε και αποτελεσματικοί στην όλη προσπάθεια. Πρώτον, πρέπει να έχουμε καλό συντονισμό μεταξύ των ρυθμίσεων αυτών και τι οδηγίε για την εξυγίαση των τραπεζών, διότι και οι δύο επηρεάζουν τον τρόπο που το επιχειρησιακό μοντέλο μπορεί να ε, μεταβληθεί εφόσον θεωρηθεί υπερβολικά περίπλοκο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να έχουμε σαφή κριτήρια που να εκφράζονται ξεκάθαρα στο νομοθεσία επίπεδο 1. Λόγω χάρη τη περιπτώσει όπου χρειάζεται διαχωρισμό ή εκεί που χρειάζονται πλέον εποπτικά μέτρα. Όλε αυτέ οι πρακτικέ λεπτομέρειε πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του επίπεδου 2. Είναι Σημαντικό λοιπόν αυτές οι δυσκολίες να ληφθούν υπόψη για να συμφωνήσουμε στο επίπεδο 1 και οι πιο περίπλοκες διαδικασίες και πολιτικές επιλογές να γίνουν και να ξεκαθαριστούν στο επίπεδο 2. Αυτός είναι ένας τομέας όπου πρέπει να έχουμε και την απαραίτητη παρακολούθηση διότι όταν υπάρξουν διαρθρωτικοί φραγμοί ε, στην αγορά θα βρεθούν τρόποι για να παρακαμφθούν. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Ευχαριστούμε κύριο Γκίγκολντ. Ευχαριστώ Ανδρέα Ένρια γιατί τονίσατε ότι εάν η ομάδα μας Άλντε βασιζόταν στην έκθεση Λίκανεν θα είχαμε καλύτερο τρόπο για να καταλήξουμε σε αυτές τις δύσκολες διαπραγματεύσεις αλλά περαιτέρω. Καλή ήταν η πρώτη πενταετία για τις εποπτικές αρχές και δε θέτε εσείς αν ορισμένα δεν μπορούν να είναι όσο καλά θα θέλαμε. Ξέρουμε πόσο περίπλοκη είναι η εποπτική δομή, δεν έχετε επαρκείς πιστώσεις, ότι έχετε νέα καθήκοντα όπως η προστασία των καταναλωτών, αλλά όχι επιπλέον προσωπικό. Και δεν φταίτε βεβαίω που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μπλοκάρει τόσο πολύ την αναθεώρηση. Ενώ το Κοινοβούλιο έχει ήδη τονίσει τα βασικά σημεία. Δεν φταίτε. Παρόλα αυτά είστε πιο ανεξάρτητοι από ό,τι θα μπορούσε κανείς να αναμένει με αυτή την δομή διακυβέρνηση. Ερωτήσεις. Πρώτον, το θέμα της αναλογικότητας στον τραπεζικό τομέα. Έχω την εντύπωση ότι εδώ μπορείτε να κάνετε περισσότερα για παράδειγμα η υποβολή εκθέσεων. Γιατί συνεχίζεται στο πλαίσιο υποβολής εκθέσεων να ζητάτε από τις τράπεζες που δεν χρησιμοποιούν το EFRS για στοιχεία που μόνο μέσω του EFRS μπορούν να τα εξαγάγουν. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Δεύτερον, ακούστηκε ότι θα υπάρξει μια τράπεζα για τον παρατραπεζικό τομέα και την επιλογή του πιο ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου. Δηλαδή θα μπορεί όποιος έχει προβλήματα να πηγαίνει σε ένα άλλο εποπτικό πλαίσιο. Θα έπρεπε να ασχοληθούν και οι τρεις εποπτικοί φορείς με αυτό και να μας προτείνουν νομοθεσία πιστεύω. Ο κύριος Ενδε... Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια κύριε Κίκολτ. Τώρα αναλογικότητα. Την ανέφερα ήδη. Θα είναι πρόκληση για μας. <clears throat> Πρέπει να εστιάσουμε πολύ εδώ την αναθεώρηση. Νομίζω ότι κάναμε μια σοβαρή προσπάθεια για να συμπεριληφθεί αυτή η αρχή σε πολλούς τομείς και στην υποβολή εκθέσεων. Υπάρχουν ε, μεγάλα τμήματα του πλαισίου υποβολής εκθέσεων που δεν αφορούν τις μικρότερες τράπεζες που εργάζονται με πιο απλό τρόπο. Να έχετε υπόψη ότι προηγουμένως ε, υπήρχε πολύ διαφορετικός όγκος στοιχείων που έπρεπε να υποβάλουν τράπεζες ανάλογα με την έδρα τους. Ορισμένες λοιπόν ε, έπρεπε να κάνουν πολύ περισσότερα από άλλες. Αλλά καταλαβαίνω τι είπατε για το IFRS. Προσπαθούμε η υποβολή εκθέσεων για τους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς να ε, παρέχουν τα στοιχεία που χρειάζονται οι εποπτικές αρχές. Ο κύριος κύριε ε, ΕΝΡΙΑ. Δεσμεύεστε ότι δεν θα επιτρέπετε στις τράπεζες, δεν θα υποχρεώνετε τις τράπεζες να υποβάλουν στοιχεία που δεν μπορούν να βγάλουν από τους λογαριασμούς τους. Η απάντησή μου είναι όχι, λέει ο κύριος Ένρια. Όχι γιατί ζητάμε από τις τράπεζες να μας δώσουν στοιχεία με ένα διαφορετικό λογιστικό πλαίσιο. Οι εποπτικές αρχές πρέπει να έχουν συγκρίσιμα στοιχεία για όλες τις τράπεζες ανεξάρτητα από το λογιστικό πλαίσιο στο οποίο εργάζονται. Φυσικά πρέπει να βασιστούμε στα στοιχεία που μας δίνουν. Αλλά πρέπει τα στοιχεία που μας δίνουν να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε ως εποπτικές. Αυτή δεν είναι λογιστική. Δεν είναι λογιστικό εγχείρημα, είναι εποπτικό εγχείρημα. Εάν είναι υπερβολικός ο φόρτος που επιβάλλουμε, μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. αλλά πρέπει να είναι αξιοποιήσιμα τα στοιχεία που μας υποβάλλουν. Από εποπτική πλευρά το χρειαζόμαστε αυτό. Για το δεύτερο σημείο που αναφέρατε, ο, τραπεζικός, ο σκιώδης τραπεζικός τομέας, η τραπεζική δραστηριότητα. Πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Και έχουμε ήδη ασχοληθεί μεταξύ των τριών αρχών. Κατά τη διάρκεια της κρίσης ε, των ομολόγων, των κρατικών ομολόγων, ε, κάνουμε προσπάθειες για να δούμε αν υπάρχει μεταφορά δραστηριοτήτων, οι τρεις ESA. Και έχουμε και την Υποπιτροπή Κινδύνων που ε, ασχολείται με αυτά ακριβώς τα θέματα. Άρα έχουμε επαρκή στοιχεία για να ε, λογοδοτήσουμε στο Κοινοβούλιο επ' αυτών. Το πρόβλημα είναι όταν οι επιχειρήσεις μετακινούνται όχι μεταξύ δικαιοδοσιών αλλά εκτός δικαιοδοσιών. Εκεί δεν βλέπουμε τίποτα. Αυτό που κάνουμε ως EBA είναι να υπάρξουν καθευτήρες γραμμές για το βαθμό στον οποίο οι τράπεζες μπορούν να εκτεθούν στον σκιώδη τραπεζικό τομέα. Μόνο έτσι μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την ε, επιλογή της κατάλληλης δικαιοδοσίας, την άγρα δικαιοδοσίας. Βέβαια είναι δύσκολο γιατί ε, πολλοί δεν μας δίνουν τα στοιχεία που θέλουμε. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλήξουμε σε αυτές τις κατευθύντηρες γραμμές, να παρακολουθήσουμε αυτές τις δραστηριότητες και να λογοδοτήσουμε σε εσά. Ευχαριστώ, ο David Coburn. Ευχαριστώ. Την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Δράγκη, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ήταν εδώ μπροστά στην Επιτροπή μας και τον ρωτήσαμε αν υπήρχε περίπτωση να ε, παρασταθεί σε μια ε, κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Η απάντησή του ήταν ότι δεν ε, ανταποκρίνεται σε διαδήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ότι και από τα εθνικά ότι ανταποκρίνεται σε τέτοια αιτήματα από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά όχι στα Εθνικά Κοινοβούλια. Τέτοιου είδους αποφάσεις λοιπόν μπορεί να επηρεάζουν τις, Ευρωπα... τις Βρετανικές τράπεζες, ε, αποφάσεις λέει, της Τράπεζας και των εποπτικών αρχών. Εάν λοιπόν σας ε, κλείτευε η Βρετανική Βουλή σε μια τέτοια επιτροπή, κύριε Ενρία, θα πηγαίνατε? Και αν ναι, τι σας διαφοροποιεί από το, σε σχέση με τον κύριο Ντράγκη, σε τι είστε διαφορετικός από τον κύριο Ντράγκη. Απάντηση. Θα απαντήσω ότι έχω ήδη παραστεί σε πολλές ακροάσεις σε εθνικά κοινοβούλια, στη Βουλή των Λόρδων, στην ε, Βουλή και την Γερουσία της Ιταλίας, αντίστοιχα στη Γερμανία, στη Γαλλία. Σε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ λοιπόν έχουν γίνει ακοράσεις, τι οποίε παρέστηνα εγώ προσωπικώ. Σε τι μπορεί να είμαι διαφορετικό, ότι έχουμε διαφορετικό ρόλο. Ρυθμιστικό και οι δράσεις τι οποίε καταλήγουμε επηρεάζουν και κανόνες που υλοποιούνται από τα εθνικά κοινοβούλια. Και χρειάζεται ως εκ τούτου ένας διάλογος και ο το, αρχικό καθήκον μας για διάλογο είναι έναντι του Κοινοβουλίου σας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι πιστεύω σκόπιμο να δίνουμε απαντήσεις και στα Εθνικά Κοινοβούλια και να εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους λάβαμε κάποιες αποφάσεις ρυθμιστικού χαρακτήρα. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Κοιτάξτε, η νομισματική πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Ο πρόεδρος κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή. Η κυρία Κάπελ, ε, εξαντλήσατε το χρόνο σας, όλοι έχουν τον ίδιο χρόνο. Μα πρόεδρε, εκπροσωπώ 4 εκατομμύρια. Εσάς ποιος σας ψήφισε. Με διακόπτετε κάθε φορά. Χωρίς μικρόφωνο. Thank you. Barbara Ευχαριστώ κύριε Κάπελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Ανδρία, θα πρέπει να επαληθεύει την λειτουργία των μεγάλων τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2016 αναδιαιτία με τη τεστ η ΕΤΑ. Πιστεύετε λοιπόν ότι μπορείτε να δώσετε μια κρίση για το βιωσιμότητα των τραπεζών και μέσα από τη διαδικασία αυτής της αξιολόγησης να επηρεάσετε και το όρια για τα ελάχιστε κεφαλαιοχικές απαιτήσει για τις τράπεζες, διότι πολλοί ανησυχούν για την ε, ε, αδυναμία, την ε, ασθενική κατάσταση του τραπεζικού τομέα, κυρίως και λόγω του τη πολιτική των πολύ χαμηλών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πιστεύετε ότι μπορείτε να αλλάξετε κάτι και βεβαίω υπάρχουν αποτελέσματα στι Ηνωμένε Πολιτείε όπου υπάρχουν ε, ιδρύματα όπω η JP Morgan που έχουν αρχίσει να δείχνουν σημαντική κερδοφορία. Έχουμε από την άλλη 25 δισεκατομμύρια ευρώ ε, κεφαλαιοχικό κενό με συνέπειες πολύ σημαντικές για τις τράπεζές μας κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας, 10.000 ε, έως το 2016 από την Barclays, 26.000 από την ε, ε, Deutsche Bank, από τη Unicredit 18.500 και άλλες. Γύρω στις 150.000 θέσεις εργασίας αναμένεται στα προσεχή χρόνια να καταργηθούν από τον τραπεζικό τομέα. Βλέπουμε χαμηλότερα έσοδα, όλο και αυξανόμενο κόστος, πίεση από τους επενδυτές στον τραπεζικό τομέα και ρωτώ κύριε Πρόεδρε την ε, ρυθμιστική αυτή πίεση που επιβάλλεται στο τραπεζικό τομέα και τις προθέσεις για όλο και περισσότερα ρυθμιστικά, ελεγκτικά, εποπτικά μέσα που θα ε, επομισθούν οι τράπεζες, πώς την κρίνεται. Ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση, γιατί έτσι μπορώ να ξεκαθαρίσω τη θέση μου για την υπερβολική ρύθμιση και την επίδραση που έχει στην πραγματική οικονομία. Νομίζω στη συζήτηση αυτή υπάρχει πάντοτε μια τεράστια παρανόηση. Αν δείτε τα δεδομένα, έχουμε δεδομένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε κράτο μέλο και αυτό που είναι σαφέ είναι ότι οι τράπεζε που δεν έχουν αρκετό κεφάλαιο λόγω χάρη, αυτέ είναι και που δανείζουν το λιγότερο. Ακριβώ διότι προσπαθούν να εξοικονομήσουν στο κεφάλαιό του και να περιορίσουν τον δανεισμό. Εάν δείτε τη διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκών Τραπεζών και Αμερικανικών, η βασική ακριβώ διαφορά είναι ότι οι Αμερικανικέ τράπεζε έχουν ε, το ε, πλεόνασμα του κεφαλαίου, ε, το έχουν φορτώσει πολύ νωρίτερα στον ισολογισμό του, έχουν εξηγιάνει και μπορούν να προχωρήσουν σε δανεισμό. Εάν θέλετε λοιπόν να παίξει δανεισμό από τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα, το πραγματικό θέμα είναι τι γίνεται με, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια λόγω της κρίσης. Έτσι θα πρέπει να δούμε τις επιλογές δανεισμού των τραπεζών. Επίσης για τον έλεγχο του κόστους και τα τεστ αντοχής. Όντως είχαμε προβολικό χρέος στην αρχή της κρίσης, οπότε ο τραπεζικός κλάδος κλείθηκε να καλύψει αυτή τη διαφορά. Σίγουρα αυτή η προβολική απέτηση πρέπει να αλλάξουμε την αναδιάρθρωση. Μόλις ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση θα είναι πιο εύρωστος ο ευρωπαϊκός ε, τραπεζικός τομέας να στηρίξει και θα είναι σε θέση να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Ευχαριστούμε κύριο Φέκμαρκ Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τις απαντήσεις σας τώρα. Να επανέλθω στο ζήτημα που φίξαμε προηγουμένως τον ασχετισμό μεταξύ διαφόρων ε, πτυχών της ενιαίας αγοράς και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι σωστό το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων. αλλά να μην υπάρχει και επικάλυψη, επανάληψη των κανόνων και των λειτουργιών. Από τη δική σας τη σκοπιά, πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπονομευθεί το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων στην ενιαία χρηματοοικονομική αγορά και πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι οι διοικητικοί πόροι χρησιμοποιούνται καταλήλως. Στο πώς θα συνδυάζετε την ε, ε, ε, δική σας προσφορά εσείς με τις άλλες αρμόδιες αρχές. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς από εδώ για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Για να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τη σωστή πολιτική ισορροπία. Αυτά είναι ζητήματα που είναι πραγματικά ουσιαστικά σημαντικά, αλλά και από πολιτικής σκοπιάς. Πώς πιστεύετε ότι να προχωρήσουμε λοιπόν στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Φατμάκη. Να προσπαθήσω να δώσω κάποια παραδείγματα, τρία συγκεκριμένα. Πρώτον, τα τεστ αντοχή. Αυτό που προσπαθήσαμε να δούμε είναι ότι τώρα προφανώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι αρμόδιες αρχές της εθνικές χώρας εκτός Ευρωζώνης να έχουν διαφορετικό πρίσμα, διαφορετική οπτική γωνία, διαφορετικούς κινδύνους, διαφορετική αντίληψη περί σχεδιασμού, όμως ο στόχος ήταν να περάσουμε από ένα τεστ αντοχής που ήταν το ίδιο για όλους όλη την ευρωπαϊκή οικονομία σε μια άσκηση αντοχής ουσιαστικά με μια κοινή μυθοδολογία ένα παρόμοιο σενάριο που ενισχύει για όλες τις τράπεζες στην ενιαία αγορά με διαφάνεια για τους επενδυτές και τους συμμετέχοντες στις τραπεζικές συναλλαγές και μετά η κάθε αρχή έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα των τεστ ε, αντοχής στις διαδικασίες δεύτερου πυλώνα για να καθορίσουν τις, για να τις κεφαλικές απαιτήσεις των τραπεζών. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη και για λόγους εποπτικών αρμοδιότητων μας ήταν σημαντικό να υπάρξει αυτή η κίνηση με κοινή μεθοδολογία και κοινέ λειτουργίες για τις χρηματαγορές. Πολύ σημαντικό για την σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η δεύτερη παρατήρηση που μπορώ να κάνω για την πολιτική, αν σκεφτούμε το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Γίνεται πολλή συζήτηση στο χώρο του ευρώ για το κατά πόσο μπορεί ένα τέτοιο πρόγραμμα να λειτουργήσει. Αλλά εφόσον υπήρχε αυτό θα έπρεπε να έχουμε κατά νου ότι αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι μια τεράστια μαζική μετατόπιση των καταθέσεων σε άλλα μέρη της ε, νέας αγοράς και μάλιστα πολλές φορές από χώρες του ευρώ σε χώρες εκτός ευρώ. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι οι καταθέτες προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την ενιαία αγορά. Αυτό είναι προφανώς αρχικά μέρος, θέμα μάλλον της Ευρωζώνης. Δεν είναι το ίδιο μια κατάθεση σε ευρώ στην Κύπρο ή στο Βερολίνο. Γιατί είναι βεβαίω θέμα του κοινού νομίσματο, αλλά είναι και θέμα τη ενιαία αγορά. Αυτή τη δική διάσταση λοιπόν πρέπει να την έχουμε υπόψη. Και το θέμα είναι επίση και η διαδικασία τη εποπτική αναθεώρηση. Έχουμε κατευθυντήρε γραμμέ για να υπάρχει κοινή μεθοδολογία μεταξύ του τι κάνει η ESSM και οι υπόλοιπε και οι κεντρικέ εθνικέ αρχέ. Είναι λοιπόν σημαντικό στις εποπτικές μας δραστηριότητε να επιλέγουμε τα σωστά ζητήματα από των οποίων μπορούμε να ε, επικεντρωθούμε και να εξασφαλίσουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εποπτών και των ε, εθνικών αρχών και εντός Ευρωζώνης και εκτός. Ευχαριστούμε κυρία Καϊλή. Thank you. Uh, so to, to follow up... Ευχαριστώ. Συνεχίζοντας ε, με βάση τις προηγούμενες ερωτήσεις θεωρείται ότι αν είναι σε καλή κατάσταση όλες οι τράπεζες, έχουν σωστούς ισολογισμούς και είναι περιορισμένη η έκθεσή τους σε κινδύνους, τότε θα είναι σε καλή κατάσταση και ο Ευρωπαϊκός Τραπεζικός Τομέας. Στην πράξη όμως διαπιστώνουμε ότι αυτή δεν είναι από μακροπροληπτική εποπτική άποψη σε συστημικό επίπεδο η καλή προσέγγιση. Χρειαζόμαστε μια ευρύτερη ε, μακροχρόνια προπτική Εάν έχουμε πιο στενή αντίληψη, τότε υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και ιδιαίτερα αναχώρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν αναχώρα προσέγγιση για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την συνολική ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα. Πώς θα πετύχουμε αυτή την ισορροπία μεταξύ μιας ευρύτερης προσέγγισης και μιας κατά περίπτωση αντιμετώπισης. Πώς αυτό αντανακλάται στη δομή των ε, τεστ αντοχής που είπατε ότι θα γίνουν το 2016 και πώς ε, θα αντιμετωπιστούν τα DTA, δηλαδή τα διάφορα στοιχεία ενεργητικού και τρίτον οι ελληνικές τράπεζες στο ελάχιστο σενάριο της ε, φερεγγιότητάς τους θεωρείται ότι είναι στο 90,5% θεωρείται στο 9,5 9,5 ναι, για, το baseline, ε, για την περίπτωση baseline θεωρείται και ότι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να ε, ε, εκτιμηθούν με τα ίδια κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Για το πώς θα εξισορροπήσουμε τα προβλήματα μεταξύ την αντιμετώπιση των προβλημάτων από συνολικό και κατά περίπτωση από συνολική κατά προοπτική, νομίζω ότι τα, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αφήνει αρκετό περιθώριο για να τα κάνουμε και τα δύο. Υπάρχει η προσαρμογή να αυξηθεί η ε, στάθμιση κινδύνου, η δυνατότητα να ζητήσουμε να αυξηθεί το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται. Έχουμε πολλή ευελιξία. Είναι σημαντικό βέβαια οι μακροπροληπτικές αρχές να εγγυηθούν ότι αυτές οι, αυτοί οι κανόνες ε, εφαρμόζονται με ενίο τρόπο. Η ιστορία μας διδάσκει ότι αν υπάρξει μια κρίση μικρών τραπεζών όπως η Κάχας στην Ισπανία μετά υπάρξει, υπάρχει επιμόλυνση και στη συνολική ευρωπαϊκή αγορά άρα πρέπει να, να τα αντιμετωπίσουμε ε, με ε, ομοιόμορφο τρόπο. Έχουμε λοιπόν την ίδια μεθοδολογία για όλα μας τα τεστ αντοχής αλλά λαμβάνουμε υπόψη και τη συμπερίληψη των ειδικών ε, κινδύνων που μπορεί να ισχύουν για κάποιες τράπεζες, σε κάποιες δικαιοδοσίες. Για παράδειγμα, φέτος έχουμε δύο κέντρα εστίασης. Ε, ο δανεισμός Forex, για την αγορά συναλλάγματος δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό στις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και τα άλλα είναι θέματα συμπεριφοράς, που και αυτό προκαλεί κινδύνους σε άλλες δικαιοδοσίες. Αυτό επιτρέπει στους επόπτες να ε, μπορούν να έχουν ε, τα αποτελέσματα από τα τεστ αντοχής τα οποία θα μας βοηθήσουν. Η ε, αντιμετώπιση των ε, αναβαλωμένων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όπως ξέρετε, η αντιμετώπιση είναι κυρίως θέμα των εθνικών αρχών. Αλλά το γεγονός ότι προτείνεται να τελειώσει για την Ευρωζώνη ε, συντομότερα αυτή η εθνική ε, δικαιοδοσία, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει να υπάρξει περισσότερο ομοιόμορφη αντιμετώπιση. Όπως είπα, δεν θα υπάρχουν κατόφλια σε αυτήν την ε, διαδικασία ελέγχου, θα είναι θέμα των εθνικών αρχών. Δηλαδή, ο SSM θα προσπαθήσει να υπάρχει συνέπεια στην αντιμετώπιση για τα κατόφλια μεταξύ όλων των δικαιοδοσιών δεν είναι θέμα κατοφλίων. Είναι κυρίως να δούμε ανατράπεζα εάν είναι επαρκές το κεφάλαιο σε σχέση με το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και τη δομή του ισολογισμού τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ανδρέα Ρία για αυτή την πολύ πλούσια ανταλλαγή απόψεων που θα αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα καλώς ορίζουμε τον κύριο Γκαμπριέλ Μπερναρντίνο. Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλιστικών και Επαγγελματικών Συντάξεων, μιας αρχής η οποία είναι προσιλωμένη στο διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας δίνω το λόγο αμέσως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Κυρίε και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ για να μοιραστώ το όραμα και τη στρατηγική μου για τον ΑΙΟΠΑ τα επόμενα χρόνια και να ανταποκριθώ ερωτήσει που θα έχετε για το ενδεχόμενο επικύρωσή μου ως ε, Προέδρου της ΕΙΟΠΑ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, το όραμά μου είναι να εξελιχθεί περαιτέρω η ΕΟΠΑ, να είναι αξιόπιστος αξιόπιστη ε, εποπτική αρχή εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου επιτήρησης. Ποιε είναι οι τρει κύριες ε, στρατηγικέ προτεραιότητε. Πρώτον, να ενισχύσουμε την ε, εποπτική σύγκληση. Δεύτερον, να ενισχύσουμε την προστασία των καναλωτών. Και τρίτον, να διατηρήσουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Πώς θα ενισχύσουμε την σύγκληση στην εποπτική δραστηριότητα με την εφαρμογή του, της οδηγίας Φεργιότητα 2 ε, θα περάσουμε από το ρυθμιστικό ρόλο στην επιτήρηση, στην εποπτεία. Και άρα πρέπει να ε, ε, περάσουμε περισσότερο στην όλο και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων. Θέλουμε να υπάρξει σύγκληση των εποπτικών δραστηριοτήτων στην Ένωση. Είναι αυτό βασικό για να εφαρμόζεται η νομοθεσία να μειωθεί η δυνατότητα επιλογής δικαιοδοσιών και να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός, θεμητός ανταγωνισμός, καθώς και το ίδιο επίπεδο προστασίας όλων όσων συμμετέχουν. Στα πλαίσια των διαφορετικών πρακτικών και νοοτροπιών μεταξύ των κρατών μελών για την υποπτική δραστηριότητα, στόχος μας θα είναι να υπάρξει περισσότερη σύγκληση προς μια ευρωπαϊκή εποπτική νοοτροπία που να βασίζεται στην εκτίμηση των κινδύνων, ούτως ώστε να υπάρχει ισχυρή αλλά δίκαιη επιτήρηση. Θεωρώ ότι η εφαρμογή του Φερικιότητα 2 είναι μια ευκαιρία προ αυτή την κατεύθυνση και θα κάνω ό,τι, μπορεί, ό,τι μπορώ για να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Στα πλαίσια αυτά, ο ΙΟΠΑ θα δώσει προτεραιότητα στη διμερή συνεργασία με τι εθνικέ αρχέ, ούτω ώστε να έχουμε ανεξάρτητη αλλά σωστή ενημέρωση για τις πρακτικές τους και να βοηθήσουμε την ε, δραστηριότητά τους ε, όπως ε, πρωτοβουλίε, όπως η επιτυχής ε, αναθεώρηση των ισολογισμών που κάναμε στη Ρουμανία και ιδιαίτερα θα ασχοληθούμε στη συνεχιζόμενη επιτήρηση και τη δημιουργία ε, σημείων αναφοράς για τα εσωτερικά πρότυπα διότι οι διαφορές εδώ μπορεί να παίξουν τεράστιο ρόλο στην διατήρηση του θεμητού ανταγωνισμού. Δεύτερον, θέλουμε να ενισχύσουμε την προληπτική προστασία των καταναλωτών. Θα το κάνουμε και από προληπτική και κατά τη διάρκεια δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Τα θέματα συμπεριφορά δεν θίγουν μόνο του καταναλωτέ, αλλά μπορεί να έχουν μια ευρύτερη προληπτική επίπτωση και μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Θα συμβάλλουμε στην ολοκλήρωση του ενιαίου εγχειριδίου για την προστασία των καταναλωτών μέσω τη εφαρμογή τη οδηγία IDD και μέσω συνέπεια σε οριζόντια θέματα, για παράδειγμα στην περίπτωση των BRIPS. Κυρίω θα ασχοληθούμε με τη σταδιακή εφαρμογή μιας ε, συντονισμένης επιτήρησης σε ενωσιακό επίπεδο με βάση τους σωστούς δείκτες και τις ε, θεματικές αναθεωρήσεις για να υπάρξει έγκαιρα ταυτοποίηση και μετριασμός των κινδύνων. Με αυτόν τον τρόπο θα επανέλθει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτή θα είναι η προστιθέμενη αξία μας. Επίσης θέλουμε να διατηρήσουμε την μακροπιστωτική σταθερότητα. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις ε, σε αυτό το τομέα. Έχουμε πολύ χαμηλά επιτόκια. Και γι' αυτό η φερεγγιότητα των ε, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ε, συνταξιωτικών ταμείων αντιμετωπίζει προβλήματα. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αξιόπιστα τεστ αντοχή για να δούμε ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι και τα τροτά σημεία και για να υπάρχουν σαφείς συστάσει για να τα αντιμετωπίσουμε με βάση το νέο εναρμονισμένο πλαίσιο για την υποβολή εκθέσεων του Φαρικιότητα 2 θα έχουμε ένα ενιαίο σύστημα για παροχή πληροφοριών ούτως ώστε να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης σε επίπεδο επιχείρησης και ευρύτερο. Έτσι θα ενισχύσουμε την ε, ποιότητα και της μικρο και της μάκρο επιτήρησης. Πέρα από αυτές τις τρεις προτεραιότητες, στα πλαίσια της εντολής μας η ΕΙΟΠΑ θα συνεχίσει να αναπτύσσει την εργασία της με βάση στοιχεία για να έχουμε μια ρωμαλαία προληπτική ε, κανονιστική ε, διαδικασία. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και τις παρενέργειες και να βασιστούμε στην ε, απλή αντιμετώπιση και την αναλογικότητα. Επειδή διαπιστώνουμε ότι συμμετέχουμε όλο και περισσότερο σε διεθνείς διοργανώσεις, θέλουμε να συμβάλλουμε περισσότερο σε διεθνείς προδιαγραφές για τον ασφαλιστικό τομέα. Και θα αναφερθώ και σε αυτά τα θέματα είμαι στη διάθεσή σας. Η ΕΙΟΠΑ θα συνεχίσει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ε, Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ούτω ώστε να συμβάλλουμε σε ένα ενιαίο προϊόν σε ευρωπαϊκή διάσταση για τις συντάξεις, το λεγόμενο ΠΕΠ μέσω σταθερών και βιώσιμων συντάξεων και επαρκών συντάξεων μπορούμε να έχουμε οικονομίες ε, κλίμακας και να βοηθήσουμε και την ε, μακροκρόνια ε, αξιόπιστη χρηματοδότηση. Και θα βοηθήσουμε αυτή τη σημαντική δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόσο ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα συμφέροντα των πολιτών έναντι των εθνικών συμφερόντων και να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα σε πλαίσιο οικονομικών, ε, οικονομικών περιορισμών και περιορισμένου προσωπικού θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε δύσκολες επιλογές. Να δώσουμε σωστή προτεραιότητα είναι πάντα αυτό πρώτο καθήκον. Η μετάβαση από τους κανόνες στην ε, εποπτεία θα πρέπει να γίνει με βάση ενισχυμένη ποιότητα στην εργασία μας. Ελπίζω να συνεχίσουμε να εργαζόμεθα σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να ανταποκρινόμεθα όσο καλύτερα μπορούμε σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Εάν με βεβαιώσετε, θα συνεχίσω να εργάζομαι ως ε, πρόεδρος της ΕΙΟΠΑ με το υψηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας, λογοδοσίας και διαφάνειας. Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσω για τις δραστηριότητές μας και τις ε, στρατηγικές μας. Για μένα η ανεξαρτησία και η λογοδοσία πηγαίνουν χέρι με χέρι. Γι' αυτό πιστεύω ότι η λογοδοσία μου έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύει την ανεξαρτησία μου προς το κοινό συμφέρον. Και προσβλέπω στη συνέχιση της προσπάθειας ε, μαζί με όλο μου το προσωπικό για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της επόμενης πενταετίας και θα συνεχίσω να εργάζομαι προς το συμφέρον των ε, πολιτών της Ένωσης και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. κύριος Βάλτς είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και κύριε Γκάμπριλ, ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση σας εδώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει προτάσεις νομοθετικών πράξεων για το Solvency 2 στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Οι συνομοθέτες έχουν καταστήσει σαφές. Πιστεύω ότι πρέπει η οδηγία να εφαρμόζεται χωρίς να ξανανοίξει όλη η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και των αναθεωρήσεων. Αλλά φαίνεται ότι να προβαίνει σε πολύ ε, ει βάθο αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη νέα τη πρόταση και με νέε ιδέε ε, για το πώ θα πρέπει να είναι αυτά τα νομοθετικά αυτής της νομοθετικής πράξης. Τι ε, βλέπετε εσείς, ποιες είναι οι θέσεις, ποιες είναι οι θέσεις της ΑΙΟΠΑ και επίσης βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια υγιή σχέση αναλογικότητας και ότι δεν τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές βάσει της εντολής ΑΙΟΠΑ. Μιλάμε για χιλιάδες ε, σελίδες εγγράφων που αποτελούν copy-paste νομοθετικών κειμένων. Βεβαίως είναι πολύ σημαντική η θέση της νομοθεσίας, πρέπει να αναλαμβάνεται δράση εκεί δηλαδή όπου έχει την συγκεκριμένη εντολή η ΟΠΑ. Μήπως θα πρέπει λοιπόν να σταματήσετε να εκδίδετε οδηγίες για το κάθε τι πώς θα ορίζατε προτεραιότητες για, τις, ε, για τα καθήκοντά σας και ποιες θα ήταν αυτές. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάλτς. Πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις σας φυσικά. Για το νομοθετικό πλαίσιο σε όλων Έχω καταστήσει σαφές και το γνωρίζετε πιστεύω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σταθερότητα στο ρυθμιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή και αντιλαμβανόμεθα βεβαίω του λόγου για του οποίου μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέλει να ρυθμίσει ορισμένα στοιχεία. Έχουμε, όπω ξέρετε, επεξεργαστεί το ζήτημα των υποδομών του τελευταίου μήνε πολύ εντατικά με προτάσεις που μπορεί να δώσουν ε, πολύ καλές και πιστικές απαντήσεις προληπτικά. Δεν μας ζητήθηκε να τοποθετηθούμε σε άλλα ζητήματα που αναπτύσσει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω πάντως όπου, ότι είναι απαραίτητο να έχουμε σταθερότητα. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να απευθύνω ένα μήνυμα ε, σύνεσης και προσοχής ως προς το να ανοίγουν πολλά θέματα. Ξέρετε ότι έχουμε δύο χρόνια μετά την ε, υλοποίηση το 2016 για την αναθεώρηση του συστήματο, όπω είπα και στι αγωγικέ μου παρατηρήσει, θέλουμε αυτό να γίνει με τρόπο διαρθρωμένο, με την αναλογικότητα, με την απλότητα ω κανόνε και εκεί πάνω σε αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε αν υπάρχει ανάγκη για νέους κανόνες. Γιατί πρέπει να αντιληφθούμε και τι συνέπειε έχουν όλα αυτά τα οποία συλλογικά ε, σχεδιάζουμε μέσα από το Solvency 2 για τα επομενα δυο 2-3 χρόνια. Και αν χρειαστούν κάποιε προσαρμογέ, τότε μόνο να γίνουν, αν διαπιστωθεί ότι χρειάζονται. Με βάση όμως στοιχεία και όχι μόνο με την ε, τάση, την έμπνευση της στιγμής σε σχέση με κάποια συγκεκριμένη πτυχή. Ε, για το άλλο ζήτημα, για την αναλογικότητα και το στοιχείο των ε, κατευθυντηριών γραμμών, θα είμαι απόλυτα σαφής κύριε Μπάλτς. Ναι, έχουμε εκδώσει μια σειρά κατευθυντηριών γραμμών. Και βεβαίω πρόκειται για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά την οποία τι εκδώσαμε. Θα συνεχίσουμε να παράγουμε κατευθυντήριε γραμμέ ε, στον αιώνα των άπαντα, γιατί τώρα μπαίνουμε στο νέο καθεστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, διότι μπορεί να μου πείτε ότι πρόκειται για χιλιάδε σελίδων, αλλά κύριε Μπάλτ, σα διαβεβαιώ ότι αν δεν υπήρχαν αυτέ οι ευρωπαϊκέ καθητήριε γραμμέ, οι χιλιάδε σελίδων που εκδώσαμε, σα διαβεβαιώ ότι θα είχαμε χιλιάδε περισσότερε σελίδε σε διεθνέ επίπεδο με αποκλίνουσες προσεγγίσεις πολύ συχνά και θα ήταν τότε πολύ πιο δύσκολο εκ των υστέρων να αποκαταστήσουμε τη σύγκληση. Γι' αυτό σας παρακαλώ να το κοιτάξετε με πολύ μεγάλη προσοχή, είναι πολύ σημαντικό. Οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε εκδώσει πιστεύω ότι όντως σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. Ξέρετε ότι, για να σας δώσω δύο παραδείγματα μόνο, αναλογικότητα σε σχέση με την απόδοση λογαριασμών. Έχουμε εκδώσει μια σειρά από ε, υποδείξεις για την απλούστευση για τις μικρότερες ε, επιχειρήσεις. Δεν χρειάζεται να δώσουν όλες τις λεπτομέρειες στις εποπτικές αρχές. Μαζί με την ΕΚΤ έχουμε συνδυαστεί για να δώσουμε οδηγίες για τις ε, αναφορές ώστε να μην γίνεται διπλή δουλειά στα στοιχεία που δίνονται στην ΕΚΤ και σε εμά. Εργαλεία, τα οποία διαθέτουμε και δωρεάν στην αγορά και ξέρω ότι πάνω από 1.200 είναι οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη που αξιοποιούν τα εργαλεία αυτά για να καλύψουν τη μετάβαση από το Solvency 1 στο Solvency 2. Είναι λοιπόν αναγκαία. Και πρέπει να σας πω, μια και προέρχομαι και από μικρή χώρα, ότι πρόκειται για, μια, ε, για μια από τις κύριες προτεραιότητες με το Solvency 2. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις αλληλένδετες. Πρώτα απ' όλα με απασχολεί το πώς θα μας επηρεάσουν τα χαμηλά επιτόκια το καλοκαίρι. Είπατε ότι οι εταιρείε ασφαλιών δέχονταν μεγάλες πίεσεις λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Και το πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης της ΕΚΤ είναι μέρη υπεύθυνο την περασμένη εβδομάδα ο διευθυντή τη ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μα είπε ότι πρόκειται να ενισχύσει το πρόγραμμα προσωπική χαλαρώση, αν ο πληθωρισμό δεν βελτιωθεί. Τι κινδύνου διαβλέπετε εσεί, Πόσο είναι ανθεκτικέ οι ε, ασφαλιστικέ εταιρείε και τα συνταξιδοτικά ταμεία, Μπορούμε να προβλέψουμε τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν, Και δεύτερη ερώτηση. Τι άποψη έχετε για την ποιότητα των τεστ αντοχής. Ένα σύστημα που ισχύει πλέον για την Ευρώπη. Ξέρουμε ότι τι προσπάθειε τη Τραπεζική Ένωση δεν έχουν επιλύθει όλα τα θέματα. Τον περασμένο χρόνο έγιναν τεστ αντοχή για τι ασφαλιστικέ εταιρείε και τώρα γίνονται για τα συνταξιδοτικά ταμεία, τα εθνικά. Τι γίνεται, υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν κενά, υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν για να βελτιωθεί το σύστημα των τεστ αντοχής τα ερχόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Δύο πολύ εύστοχε ερωτήσει και όπως είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία Θέλουμε να διαβεβαιωθούμε ότι υπάρχει σταθερότητα και των συνταξιδοτικών και των ασφαλιστικών και αυτό βεβαίω είναι προτεραιότητα από τι πρώτε για το μέλλον. Για την χαμηλή κερδοφορία και την επιρροή του προσωπικής χαλάρωση είναι σαφέ και είναι κοινώ γνωστό ότι σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που τα μέτρα μακροοικονομικής νομισματικής πολιτικής το ενισχύουν, δημιουργεί σοβαρότατες προκλήσεις στον τομέα των ε, ασφαλίσεων. Γι' αυτό επικεντρωνόμαστε ω προστατέστα αντοχής σε αυτές ακριβώς του κινδύνους. Διότι εάν δει κανεί τι γίνεται από τη σκοπιά των συντάξεων και των ασφαλίσεων, το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων όχι μόνο αυξάνει τον, ε, τους σοβαρότητα του παθητικού, αλλά δεν, αυξίζουν, δεν αυξάνονται τα, ενεργητικά στοιχεία, τα στοιχεία του ενεργητικού με τον ίδιο τρόπο που αυξάνονται αυτά του παθητικού. Οπότε, για λόγους φερεγγιότητας, τελικά καταλήγει κανείς να συνειδητοποιείται και λιγότερη κερδοφορία. Αυτό είναι ένα θέμα το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά ως αποτέλεσμα των τεστ αντοχής έχουμε δώσει σαφείς συστάσεις στις εθνικές αρχές ώστε να εξετάσουν που τα ε, ε, μοντέλα, η δομή που έχει δημιουργηθεί ε, έχει προβλήματα. Και αυτό ισχύει κυρίως όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην εξισορρόπηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Όταν εκεί υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν και προβλήματα με τις επανεπενδύσεις. Και μετά από ένα-δύο χρόνια είναι λίγο δύσκολα, αλλά μπορεί να προκύψουν ακόμη και προβλήματα ροής ε, μετρητού. Περιμένουμε λοιπόν αυτά να μην πάρουν ε, μια τέτοια μορφή που να μην αλλάζει πλέον, αλλά να παρέμβουμε γέρο. Να αλλάξουν οι εταιρείε το τι τους προϊόντα προσφέρουν, να δουν αν έχουν επιβάλει τις ε, διατάξει που ισχύουν. Αυτό από ό,τι προβλέπουμε με το Solvency 2 θα συμβεί αργά ή γρήγορα. Οπότε και οι εταιρείε που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο θα πρέπει να ενισχύσουν βήμα-βήμα την ε, κατάσταση τη φραγκιότητά του ω προ την ποιότητα των τεστ αντοχή. Τα τεστ αντοχή που κάνουμε πιστεύουμε ότι είναι αξιόπιστα. Προσπαθούμε να ε, εντείνουμε το επίπεδο πληροφοριών που παρέχουμε εκτός. Ε, αυτό θα μα φέρει και το Solvency 2 περισσότερη διαφάνεια, αλλά ως προς την ποιότητα του τεστ. Ένα-δυο σχόλια να κάνω. Θα θέλαμε να μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα τα ίδια τα τεστ αντοχής. Ακόμα εξαρτώμαθα υπερβολικά από τις εθνικές αρχές. Δεν μιλούμε απευθεία με τους ε, ασφαλιστικούς ομίλους, μιλούμε μέσω των εθνικών αρχών και αυτό μας δυσκολεύει. Μας δυσκολεύει για να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε ε, σίγουροι για τα αποτελέσματά μας. Αυτό πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστούμε κυρία Σούιμπαν. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους, διότι οι ερωτήσεις μου στους τρεις διαφορετικούς υποψηφίους έχουν, έχουν μια συνέχεια μεταξύ τους. Για του κανόνε τη περασμένη θητείας, λοιπόν, όπω αναφέρθηκε και προηγουμένω, θα ήθελα και στη δική σας ομάδα να απευθύνω επένους για το πώς χειριστήκατε όλα αυτά που προέκυψαν από την πρώτη θητεία, από την προηγούμενη θητεία και τις κατευθυντήριε γραμμές σας. Όμως, όπως θα προχωρούμε στις προτεραιότητέ μας, θα χρειαστούμε και άλλα εργαλεία. Ε, όχι απλώς την πλήρη ολοποίηση, αλλά την επιβολή των ε, κανόνων του ενιαίου χειριτή από τις αρμόδιες αρχές. Τι θα κάνετε λοιπόν με τα έγγραφα τα απαντήσεων. Πώς θα εξασφαλίσετε διαφάνεια για τους συνομιλητές σας, ιδίως ε, στο πώς θα καθορίσετε την ε, πορεία ε, για το μέλλον και πώς θα συνεννοηθείτε με το Ευρωκοινοβούλιο όταν θα ετοιμάζετε τα έγγραφα για τη, των ερωταπαντήσεων για, τους, για τις αρμόδιες αρχές και τις και τους ενεργοποιούμενους στην αγορά. Επίσης, τι μέτρα μπορείτε να πάρετε στο επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου σας για να βεβαιωθείτε ότι θα έχετε πλήρη εφαρμογή των κανόνων του επίπεδου 1. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σουίνμπεν. Ε, πολύ καλές ερωτήσεις. Νομίζω ότι βρισκόμαστε περίπου στην ίδια θέση, όπως είπατε, και έχουμε τον ίδιο στόχο για ε, την εποπτεία, λοιπόν. Και αυτό που είπατε ε, για τα ερχόμενα χρόνια σαφώς είναι προτεραιότητα και τώρα ε, για το ενιαίο εγχειρίδιο και για να υπάρχει συνέπεια στην εφαρμογή των αποκτικών αρχών. Βεβαίω, οι κατευθυντήριε γραμμέ μα είναι ένα θεμελιώδη στοιχείο για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν σαφεί ενδείξει προ τι αρχέ και τι εταιρείε για το πώ να εφαρμόσουν το όλο σύστημα. Έπειτα με τη διαδικασία εξέτασης οποτήμων, αυτό ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο και θα, θα συνεχίσει. Όμως έχουμε και μια σειρά από άλλα εργαλεία από το καταστατικό μας και μπορούμε να τα προωθήσουμε. Λόγου χάρη έχουμε μια ομάδα ε, επισκόπησης της εποπτείας. Ε, για έχουμε μόνο τέσσερις συνεργάτες σε αυτή την ομάδα, δεν έχουμε προπολογισμό για κάτι καλύτερο προς στιγμή αλλά αυτοί οι άνθρωποι συναντούν του εκπροσώπους των εθνικών αρχών και κοιτάζουν πώ το όλο σύστημα θα εφαρμοστεί. Βλέπουν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τι επιμέρου αγορέ, όχι μόνο προ την συνοχή, αλλά και την ποιότητα των διαδικασιών αποκτία. Να είμαι πολύ σαφή. Μπορεί να λέμε ότι έχουμε ενιαία εσωτερική αγορά. Εάν όμω δεν έχουμε διαρκή εποπτεία και βαριέ επίπεδο δεν θα έχουμε ποτέ εσωτερική αγορά. Και το πρόβλημα είναι ότι τώρα έχουμε διαφορετικά επίπεδα εποπτείας στην Ευρώπη. Ε, αυτό λοιπόν το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά και πρόσφατα κάναμε μια προσπάθεια σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές με πολύ διαφανή τρόπο ε, να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα σε μια μελέτη για το πώς εφαρμόζουν οι εταιρείε τους κανόνες του Solvency 1 και 2 με τις κεφαλικές απαιτήσει είδαμε που αν λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ανεπάρκειες γιατί χρειάζεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο ε, επιβολής των κανόνων για να μπορέσει να έχει, να μπορέσει να έχει εμπιστοσύνη η αγορά. Αυτό θα πρέπει να δούμε στο μέλλον, να υπάρχει ποιοτικό ρόλο εποπτείας. Ευχαριστούμε κυρία Γκουλά. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και εγώ θα έχω μια συνέχεια στις ε, ερωτήσεις μου. Ανησυχώ για τη σχέση μεταξύ του επίπεδου 1 και των άλλων κανόνων. Θεωρώ ότι έναντι της κοινή γνώμης δεν πρέπει να υποτιμήσουμε. Σε τι βαθμό όλη αυτή η πληθώρα κειμένων δημιουργεί σύγχυση. Βεβαίως, είναι πρόσφατα αυτά τα όργανα, αλλά αυτή η σύγχυση θίγει την εικόνα της Ευρώπης σκοπεύετε να μειώσετε σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των κατευθυντηρίων γραμμών και να μην προβλέπετε αποφάσεις που θα ληφθούν. Και δεύτερον, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε ούτως ώστε να υπάρχει μια συνεκτικότητα μεταξύ αυτών που συμβαίνουν σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρετε ότι το FSB ασχολήθηκε με τον ασφαλιστικό τομέα, τι μπορούμε να κάνουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Για το πρώτο θέμα, για τα επίπεδα 1, 2, 3. Κοιτάξτε. Θέλαμε η οδηγία μας για την φερεγκαιότητα να βασίζεται σε αρχές, αλλά ο διάβολος είναι πάντα στις λεπτομέρειες. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα στο φερεγκαιότητα 1 που είτε δεν επελήθησαν είτε αντιμετωπίστηκαν με αρκετά ασαφείς συμβιβασμούς που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην πράξη και στα επίπεδα 2 και 3 φυσικά πρέπει να υπάρξει περισσότερη λεπτομέρεια. Συνολικά θα έλεγα ότι όλοι θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν στο επίπεδο 1 να λύσουμε τα πάντα, να υπάρχουν όλες λεπτομέρειες, γιατί θα ήταν τότε υπερβολικά περιοριστικό. Και ξέρετε βέβαια η κατάσταση στην αγορά επίσης κινείται. Πρέπει και εμείς να μπορούμε να αλλάξουμε την αντιμετώπιση μας. Θεωρώ λοιπόν ότι ο καλύτερος τρόπος θα είναι σε επίπεδο ένα να αναφερόμεθα στις αρχές και κατόπιν να δίνουμε στα άλλα επίπεδα με κάθε λογοδοσία προς το Κοινοβούλιο και τους άλλους περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειε. Αυτός νομίζω θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα για τα διεθνή πρότυπα τα συζητάμε. Στον ασφαλιστικό τομέα, ευτυχώς από τότε που ξεκίνησε ο ΕΙΟΠΑ, υπήρξε συμφωνία στο Συμβούλιο μας ότι θα συμμετείχαμε στη διεθνή συναντήση στο IIIS. Νομίζω ότι είναι αρκετά συντονισμένη η προσέγγιση μας και η στάση μας έναντι του IIIS. Εκεί που υπάρχει ένα κενό έχει να κάνει με το FSB, γιατί δεν συμμετέχουμε εκεί το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Δεν ε, ενημερωνόμεθα. Η εργασία για, την, ε, για τα νομοθετήματα για την εξυγίανση και ανάκαμψη συνεχίζεται. Ε, νομίζω ότι καλό είναι να καταλήξουμε πριν υπάρξει τελική απόφαση, γιατί εδώ ακριβώς έχουμε ένα κενό. Ευχαριστώ, είναι όντως θέμα, λέει ο Πρόεδρος. Ο Σβέν Γκίγκολτ. Καλώς ήρθατε και πάλι. Όπως βλέπω εγώ, όπως βλέπουμε εμείς τα πράγματα, επιδεικνύεται πολύ θάρρος. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχατε νομική βάση για τις δράσεις σας. Γιατί υπάρχουν συστημικοί κίνδυνοι στον κλάδο των ασφαλίσεων και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσετε τη δράση σας βεβαίως με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Έχουμε κάνει πολλές περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε την ε, ρύθμιση του τραπεζικού τομέα σε σχέση με, αυτή, με την ρύθμιση του ασφαλιστικού. Δεν βλέπουμε δηλαδή να είναι προσαρμοσμένο το κανονιστικό πλαίσιο για τον ασφαλιστικό τομέα στις εξελίξεις που θα δούμε να συμβαίνουν στον τραπεζοπιστικό τομέα. Άρα και ενώ παίρνω όλο και πιο πολλούς, αναλαμβάνω όλο και πιο πολλούς κινδύνους οι ασφαλίσεις. Εσείς θα δώσετε προτάσεις προς τους συνομοθέτες για την αναζήτηση της πιο ευνοϊκής δικαιοδοσίας και άλλες προτάσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη μιας εκθέσεως σχετικής με αυτό το κίνδυνο και τη σκιώδη τραπεζική δραστηριότητα βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ Σβέν από τελευταία παρατήρηση, ο ορισμός της κοιόδους τραπεζικής δραστηριότητας είναι κάπως σαφής όπως ξέρετε. Για μας, όταν μιλούμε παραδείγματι ε, για παρέμβαση των ασφαλιστικών ε, ταμείων σε δραστηριότητες δανειοδοτικές, για μας δεν είναι, τραπεζική, δεν είναι σκιώδης τραπεζική δραστηριότητα. Είναι, γιατί είναι πολύ συνηθισμένο αυτό, είναι μια δευτερογενής δραστηριότητα, πολύ περιορισμένη, 1% και λιγότερο των, του ενεργητικού, των ασφαλιστικών, με διαφορά εκτός από, το, από τις κάτω χώρες ε, και την Γερμανία, όπου είναι πολύ πιο υψηλά τα ποσοστά για λόγους νομοθετικούς και διαμόρφωσης του ε, συστήματος. Άρα λοιπόν, αυτό που βλέπουμε τώρα δεν σημαίνει μία ριζική αλλαγή. Βλέπουμε επενδύσεις βέβαια για τις υποδομές, για συγκεκριμένες επενδύσεις και το παρακολουθούμε μαζί με τους αδέλφους της ε, Κοινής Επιτροπής. Διαρκώς το παρακολουθούμε και με την εισαγωγή του ΟΡΜΑΝΣΗ 2 θα έχουμε πολύ καλύτερες πληροφορίες στη θέση μας για να αναλύσουμε τα ζητήματα αυτά της υλοποίησης και βέβαια να επικεντρωθούμε και, σε, και συγκέντρωσης μάλλον κινδύνων σε συγκεκριμένου τομεί. Αλλά α μην μιλούμε για σκιώδη τραπεζική δραστηριότητα ελαφρά την καρδία, γιατί όπω είπε και νωρίτερα ο συνάδελφο είναι ζητήματα που γίνονται χάρη γίνονται όταν δεν υπάρχουν ρυθμιστικές βάσεις. Θα κοιτάξουμε το Solvency 2 εάν υπάρχει ζήτημα ε, προτίμησης δικαιοδοσίας και εάν θα πρέπει να παρέχουμε και βεβαίως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνονται τις δραστηριότητες ε, θα κοιτάξουμε αν έχουν τις κατάλληλες δυνατότητες ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου. Αυτό θα το κοιτάξουμε, η δουλειά μας ως αποπτικών αρχών. Ευχαριστώ, Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικές ερωτήσεις, διότι είμαι ο εισηγητής της ομάδας μου για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ΕΟΠΑ. Όταν ε, είναι χαμηλά τα επιτόκια, μερικοί αναζητούν κέρδη και από παράγωγα που μπορεί να είναι επικίνδυνα, αρκετά διακειμενόμενα και δεν έχουν και μεγάλη ρευστότητα. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί τα ασφαλιστικά να κάνουν και επενδύσεις πολύ επιθετικές. Οπότε αυτό που διερωτώ είναι εάν είστε υπέρ της πολύ συγκεκριμένου, πολύ περιορισμού τέτοιων εργαλείων. Ή λέτε ότι καλύτερα είναι να έχουμε συντηρητική στάση. Το πρόβλημα είναι μήπως από μία μικρή σπίθα ε, τελικά καταλήξει να ε, μην υπάρχει επαρκής προστασία των ε, αποταμιεύσεων των εργαζομένων. Είπατε επίσης ότι να υπάρχουν σωστά ε, θεμέλια στην ε, υποδομή είναι καθοριστικό για την οικονομική ανάπτυξη και να υπάρξουν επαρκείς επενδύσεις, το ίδιο και για τα συνταξιδοτικά ταμεία λοιπόν. Ε, τι κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας προτείνεται. Βλέπουμε ότι κάποιες φορές η δομή στο project financing δεν φέρνει αρκετό κέρδο για τους επενδυτές μιλάμε για επενδύσεις, ιδιαίτερα επικίνδυνες με μεγάλο ποσοστό κινδύνου. Τι οικονομική βιωσιμότητα λοιπόν ε, βλέπετε και μια τρίτη παρατήρηση. Με συγχωρείτε, αλλά φτάσατε τα δύο λεπτά. Ευχαριστώ για τις διερωτήσεις σας. Ε, πρώτα απ' όλα για τα συντεξοδοτικά και τις επενδύσεις τους. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή το ρυθμιστικό περιβάλλον στην Ευρώπη για τα συνταξιδοτικά είναι αρκετά μινιμαλιστικό για τον όγκο κανόνων που υπάρχουν. Έχουν τεράστια ευελιξία τα κατημέλη για το πώ θα εφαρμόσουν αυτέ τι οδηγίε και στον τομέα των επενδύσεων. Ε, κάποιο θα πρέπει απλώ να είναι συνετό. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει στο επίπεδο των κρατών. Είναι βεβαίω δύσκολο για μα να ε, εξασφαλίσουμε περισσότερη συνοχή σε αυτό το τομέα. Είδα ότι κάθε, κάθε μέλο έχει του δικού του ιδιαίτερου κανόνε. Από τη δική μου την ε, σκοπιά και ω προ τι επενδύσει των συνταξιδοτικών ταμείων, είναι σημαντικό βεβαίω να έχουν κατά καλή διαχείριση του ενεργητικού του του στα συνταξιωτικά, διότι αυτό εν τέλει θα του προσφέρει τη δυνατότητα να έχουν ε, και απόδοση για, τους, για τα μέλη του, του συνταξιούχου. Έχουν όμως και κάποια δάνεια ε, μακροχρόνια, οπότε εκεί κάτι πρέπει να γίνει, γιατί οι μακροχρόνιες επενδύσεις τότε αποκτούν νόημα. Όμως εξαρτάται και τι υπόσχεση σύνταξη δίνει κανείς. Διότι αν ένα συνταξιωτικό πρόγραμμα έχει μεγάλη ρευστότητα, δηλαδή μπορεί κανείς να πάρει τα χρήματα ανά πάσα στιγμή, δεν μιλάμε για ένα προϊόν συνταξιδοτικό. Δεν μπορεί κανεί να επενδύσει τόσο μακροπρόθεσμα, διότι θα αντιμετωπίσει, θα προσκρούσε στους υφάλου τη ρευστότητα. Είναι λοιπόν ένα θέμα εξισορρόπησης ενεργητικού και παθητικού. Για τα θέματα υποδομών στην ΕΟΠΑ κάναμε μία μελέτη και καταλήξαμε στο εξή συμπέρασμα για τη νέα ε, κατηγορία αυτή στοιχείων του ενεργητικού και τη σύνθεσή τους. Δεν μιλάμε για οποιοδήποτε ε, είδους ε, υποδομή, αλλά για κάποιο είδους μόνο σύνθεση του ενεργητικού με τις ροές μετρητών, με τα τεστ αντοχής Αυτό που θελήσαμε είναι να δούμε ότι στα Εδώ πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει αντιμετώπιση σωστή αυτού του παράγοντα κινδύνου στο project financing. Και μετά για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά καλά ε, ε, έργα εδώ ε, τα προγράμματα έργων τα αναλαμβάνουν οι μεγαλύτερε εταιρείε που έχουν ε, και την περισσότερη ισχύ στην αγορά και κάνουν γρήγορα τη σωστή ανάλυση. Μικρότερε και πιο περιορισμένε θα έχουν τα λιγότερο ποιοτικά έργα. Οπότε πρέπει να έχουν πολύ μεγάλε δυνατότητε αντιμετώπιση του κινδύνου για να τα ε, φέρουν ει πέρα. Αυτό θέλουμε να γίνει με βιώσιμο τρόπο στην όλη μα προσπάθεια. Αυτό επιδιώκουμε. Ευχαριστούμε ο κ. Σάνεμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ απλή η ερώτησή μου. Ως ένας απλός άνθρωπος σε αυτή τη συνάντηση εμπειρογνωμόνων έχω κάθε σεβασμό για το φορέα σας γιατί ασχολείστε με την ε, σταθερότητα των συντάξεων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ο ρόλος σας είναι σημαντικός και σας εκτιμούμε. Ο κύριος Ντράγκη ήταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν ιδιαίτερα λακωνικός. Είπε ότι η σταθερότητα και η κερδοφορία δεν είναι βασικό και κεντρικό καθήκον της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια συστημικών κινδύνων και παρέμπεψε σε αυτήν. Και το ρώτησα ότι η πολιτική επιτοκίων της ε, ΕΚΤΑΦ δεν δημιουργεί συστημικούς κινδύνους. Επειδή λοιπόν ήταν τόσο σύντομος, επειδή είχε πει ότι δεν ήταν ευθύνη του, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο γιατί νομίζω ότι η πολιτική επιτοκίων ε, προκαλεί ε, μεγάλους κινδύνους για το δικό σας θεσμικό όργανο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Βεβαίω το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά από την αρχή ήδη το 2011 όταν ξεκινήσαμε. Δημοσιεύσαμε μια γνώμη για τις επιπτώσεις των χαμηλών επιτοκίων και την αποστήλαμε στην ε, Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου. Νομίζω ότι η κατανόηση των επιπτώσεων της ε, νομισματικής πολιτικής και των χαμηλών επιτοκίων αυξάνεται και η ΟΠΑ συμμετέχει στη συζήτηση. Έχουμε μια ομάδα που συζητάει την επίπτωση των χαμηλών επιτοκίων όχι μόνο στην οικονομία αλλά και σε άλλους τομείς πέραν του τραπεζικού τομέα, ιδιαίτερα λοιπόν στον ασφαλιστικό τομέα και στον τομέα των συντάξεων της ποσοτικής χαλάρωσης. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ στην κατανόηση των επιπτώσεων αυτών των ε, ενεργειών. Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα από μια σταθεροποίηση της οικονομίας θα επωφεληθούν και οι ασφαλιστικές ε, εταιρείες και τα συντοξιωτικά ταμεία. Το πρόβλημα όμως είναι στην πορεία προς αυτό. Και όσο περισσότερο κρατάει αυτή η περίοδος τόσο χαμηλών επιτοκίων, τόσο περισσότερο θα είναι οι επιπτώσεις. Κάνουμε λοιπόν ότι μπορούμε από πλευρά μας με πολύ διαφανή πιστεύω τρόπο και ίσως μπορούμε να πούμε και κάποιες φορές ανδρείο τρόπο. Βεβαίως είμαστε στη Φραγκφούρδη, οπότε είμαστε συνεχώς σε διάλογο με την ΕΚΤ και φυσικά και προσωπικά με τον Μάριο τα πάμε πολύ καλά. Ο Βέρναρ Λάνιαν. Ευχαριστώ κύριε Βερναρντίνο. Πολλές φορές έχετε τοποθετηθεί εδώ στο Κοινοβούλιο για τις ε, προτάσεις που έχετε δημοσιεύσει. Δεν εγκρίναμε την, ε, το αίτημά σας για ενίσχυση του προπολογισμού. Ίσως θα έπρεπε να αναστηθούν και τα αίτια, γιατί μπορεί τα αίτια να έγκυνται στο ότι ανέλαβε πρωτοβουλίες η ΕΙΟΠΑ στο παρελθόν που δεν καλύπτονται από την νομοθεσία επίπεδου 1, δηλαδή ανέλαβε δικές της πρωτοβουλίες με πολλές οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές καλύτερα, του Solvency 2 και με εξουδοξής και ε, επίσης 672 δράσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Καλή βέβαια είναι η ίδια πρωτοβουλία, αλλά βλέπω να ε, μας απειλεί μαζική υπερβολική ρυθμιστική δραστηριότητα στον ασφαλιστικό τομέα. Λέτε ότι θέλετε να προβάλλετε καλές λύσεις. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να προβάλλετε τις λύσεις που έχει επιλέξει ο νομοθέτης. Και στη συζήτηση για την διαμεσολάβηση στην, στον ασφαλιστικό τομέα. Θέλω να σας επισημάνω τα εξής. Έχουμε το εγχειρίδιο ενημέρωσης για τα προϊόντα που θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή 12 μήνες μετά την έγκριση των προδιαγραφών το έχουμε συζητήσει και επεξεργαστεί και δεύτερον την ένταση με την οποία ε, προχωρεί στις ε, προδιαγραφές της για τα προϊόντα στο άρθρο 1α παρότι ε, είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το σύστημα των κατεξουδότηση πράξεων να εκδίδει τις σχετικές οδηγίες. Άρα ρωτώ, έχετε ξεπεράσει κάποια όρια αρμοδιοτήτων και μήπως μακροπρόθεσμα αυτό σημαίνει και αλλαγές στην, και επίδραση μάλλον στην πολιτική των χαμηλών επιτοκίων. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκεν. Θα εστιαστούμε σε δύο κύρια ζητήματα νομίζω. Καταρχάς τις ίδιες πρωτοβουλίες. Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε. Σας διαβεβαιώ ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε απορρέουν 100% από όσα προβλέπει η εφαρμοζόμενη σε εμά νομοθεσία, σε κάθε τομέα. Μπορεί να συμφωνεί κανεί να διαφωνεί με τον αριθμό των κατευθυντηρίων γραμμών που εκδίδουμε. Όπω απάντησα όμω και νωρίτερα στον κύριο Μπάλτ, πιστεύω ότι αυτό που πράττουμε είναι προ το συμφέρον γενικά της ε, ισχνότητας τη ε, νομοθεσία, γιατί διαφορετικά θα είχαμε αντικρουόμενες κατευθυντήρες γραμμές σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, σε σχέση με ένα τεστ αντοχή για τον ασφαλιστικό τομέα που αμφισβητήθηκε σαν να μην είχαμε τη δυνατότητα εμεί από την νομοθεσία που, μας, που ισχύει στον τομέα μας να προβούμε σε τεστ αντοχή των ασφαλιστικών ε, ταμείων. Κοιτάξτε, προφανώ και το έχουμε και ό,τι κάνουμε έχει να στηρίζεται στην νομοθεσία μα είμαι απόλυτα σαφή σε αυτό. Είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για την εφαρμογή της οδηγίας το IDD δηλαδή, βεβαίως και θα δώσουμε ευρωτερότητα σε αυτό, η προστασία του καταναλωτή είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία των στρατηγικής μας. Θα αναπτύξουμε αυτό το ε, εγχειρίδιο ενημέρωσης που προβλέπεται από την νομοθεσία, που ξέρουμε επίσης ότι υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως ε, επεξεργαζόμαστε ζητήματα εποπτείας προϊόντων και διακυβέρνησης, ζητήματα που ε, περιλάβαμε σε διαβουλεύσεις μας τις λεγόμενες προπαρασκευαστικές καταστηρίες γραμμές. Με βασική ιδέα την εξής, ότι όταν ε, οι αρχές εποπτείας των κρατών μελών και οι επιχειρήσεις αρχίζουν να εφαρμόσουν το ενημερωτικό αυτό φυλάδιο, το ITD, το κάνουν με βάση κάποιες ε, κοινέ αρχές, όχι ο καθένας από την πλευρά του, ώστε στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τη σύγκληση και όπω κάναμε και με το Solvency 2. Εκδώσαμε το 2014 κατευθυντήριε γραμμέ και αφήσαμε δύο χρόνια προετοιμασία για το Solvency 2. Και νομίζω ήταν καλή επιλογή αυτή. Διότι τώρα έχουμε αυτή την ε, συνοχή στην προετοιμασία για την ε, θέση εφαρμογή του Solvency 2. Πολύ καλύτερα από ότι αν δεν είχαμε κάνει τίποτα, αν δεν είχαμε δώσει τι τις γραμμέ. Αυτή είναι η επιλογή μα. Και κύριε Λάγκεν, προτεραιότητες ορίζουμε κάθε μέρα. Προφανώς και είναι η δουλειά μας. Και θα ορίζουμε ε, προτεραιότητες όπως είναι αυτές απαραίτητες για να κάνουμε στο τη δουλειά μας, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Γκέλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η αγορά, η ένωση κεφάλαια αγορών είναι μια μεγάλη προτεραιότητα και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα συνταξιδευτικά μάλλον, είναι μεγαλύτεροι επενδυτέ εδώ. Θα έχουν ζωτικό ρόλο στην εφαρμογή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση τη Επιτροπή ενθαρρύνει του επενδυτέ να επενδύουν σε τίτλου ώστε να ε, αντιληφθεί περισσότερο κεφάλαιο στην πραγματική οικονομία. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές ε, επιφυλάξεις για το κατά πόσο έτσι θα χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες και κατά πόσον ε, είναι δαπανηρό αυτό και δεν θα υπάρχει δυνατότητα σωστής παρακολούθησης. Ε, αυτό που με απασχολεί είναι το κατά πόσο έχετε ανάλογες ανησυχίες, το κατά πόσο η τυπλοποίηση θα είναι ένα σωστό εργαλείο για ε, να χρηματοδοτούνται και οι μικρομεσαίες και πώς αντιμετωπίσετε το συστημικό κίνδυνο. Και μια πολύ σύντομη ακόμη ερώτηση. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες. Πολλοί από τους προφόρους μου ήρθαν και με ρώτησαν και μου είπαν ότι οι ασφαλιστικές ε, είναι πολύ άνετες με το θέμα της, του απόρριτου του, των προσωπικών δεδομένων. Τα χρησιμοποιούν πολλές φορές για εμπορικού σκοπούς. Τι θα κάνετε λοιπόν για να βεβαιωθείτε ότι οι ασφαλιστικές δεν μεταφέρουν δεδομένα για επορικούς σκοπούς. Σας ευχαριστώ. Πολύ καλές και δυο σας ερωτήσεις για την τυπλοποίηση. Το είδαμε και πριν από δύο χρόνια νομίζω, στα πλαίσια του Solvency 2, με το σκοπό να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ της αποδοτικής τυπλοποίησης και της μη αποδοτικής. Είδαμε ότι υπήρχαν διαφορετικέ συμπεριφορέ και διαφορετικέ αποδόσει από άλλα είδη ε, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Οπότε κάποια στιγμή καταλήξαμε σε κάποιε συστάσει ε, και συστήσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μια τέτοια προσέγγιση με ψηλή ποιότητα τυπλοποίηση και χαμηλότερη βέβαια, αλλά να γίνεται σωστή διαφοροποίηση από την προληπτική σκοπιά. Αυτό νομίζω ότι είναι το σωστό που πρέπει να κάνει μέσα σε κάθε περίπτωση. Διότι είναι διαφορετική κίνδυνη ανάλογα με τα τυπλοποίηση. Πώ μπορούμε να τα βελτιώσουμε αυτά, πρέπει να συνεργαστούμε με του συναδέλφου μα τη EVA για την ε, ενιαία διαφανή τυπλοποίηση με στοιχεία που νομίζω ότι αν το πετύχουμε θα είναι θετικά. Για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και για αυτή την αγορά και για να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τους επενδυτές και τους ασφαλιστές. Θα είναι νομίζω η σωστή, το σωστό βήμα στην κατεύθυνση η διπλοποίηση και καλά να γίνεται, αλλά και να λαμβάνονται υπόψη είναι κίνδυνοι. Να μην γίνονται ανεξέλεγκτα αποδεκτά κάποια πράγματα και φτάσουμε σε καταστάσεις του παρελθόντος για την τυπλοποίηση τώρα. Για το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων, ο τομέα των ασφαλιστών αυτή τη στιγμή ε, αντιμετωπίζει μια τεράστια αλλαγή λόγω της ψηφιοποίησης των πάντων. Τα μεγάλα δεδομένα, όπως αναφέρονται επίσης, είναι ένα θέμα. Ε, αυτό το βλέπουμε από τη σκοπιά του καταναλωτή βεβαίω. Και το έχουμε υπόψη στο πρόγραμμα της Μικρής Επιτροπής για το 2016 αλλά βλέπουμε πολύ προσεκτικά πώς τα δεδομένα τα αντιμετωπίζουν οι διάφοροι τομείς, οι επιμέρους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο ασφαλιστικός. Θα επανέλθουμε εδώ, διότι δεν θέλουμε να ανακόψουμε την καινοτομία με ένα, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι για τους καταναλωτές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γκάμπριελ, για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Ήταν πολύ καλή αυτή η ευκαιρία να τα συζητήσουμε μετά την τόσο θετική εμπειρία που είχαμε στην πρώτη συστητία. Ευχαριστώ. And now... Steven Major. Ε, τώρα ο κύριος Steven Major ο πλευρά της ΕΣΜΑ, πρόεδρος της ΕΣΜΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Ευχαριστώ Ρομπέρτο για αυτή τη σύντομη σύσταση. Ε, μέλη του Κοινοβουλίου κυρίες και κύριοι. Ταξίδευσα σήμερα από το Παρίσι, όπου ξέρετε έχει την έδρα της ΕΣΜΑ. Όπως όλοι ε, είμαστε, είμαι σοκαρισμένος και νιώθω μεγάλη θλίψη για τη γεγονότα της Παρασκευής. Το Παρίσι είναι πια το σπίτι της ΕΣΜΑ τα τελευταία χρόνια. Είναι μια χώρα, μια πόλη για την οποία έχουμε έντονα αισθήματα. Έχουμε λοιπόν στέλνουμε τις σκέψεις μας στα θύματα και όσους έχασαν τους αγαπημένους μας και πραγματικά θα είμαστε σταθεροί στο, στη στήριξή μας για το Παρίσι και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε πέραν αυτών πρέπει να πω ότι ε, αυτή την αναστάτωση, ε, την, ε, πέρα από την αναστάτωση, πρέπει να πω για το, στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ ότι είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκουμε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε την παράταση της θητείας μου. Εφόσον ανανεωθεί η θητεία μου θα μπορέσω να συνεχίσω αυτή την εξαιρετική εμπειρία να έχω υπάρξει πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΣΜΑ. Από τη στιγμή της ίδρυσης της ε, η ΕΣΜΑ έχει αναλάβει ένα μεγάλο φάσμα αρμοδιοτήτων με περιορισμένους πόρους. Όλα έχουν συμβάλει στους τρεις βασικούς ε, στόχους της προστασίας των επενδυτών, της ευρωτικής των αγορών και της θεματοποιητικής σταθερότητας. Έχουμε συμβάλει τα μάλλα στην καλή λειτουργία των ε, ευρωπαϊκών χρηματαγορών που είναι ο ακρογωνής λίθος της οικονομικής ανάπτυξης. Αν κοιτάξουμε προς το παρελθόν, η ίδρυση της ΕΣΜΑ από το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν μια αλλαγή αλλαγή Καμπή, ε, ένα ορόσημο που νομίζω ότι πέτυχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είχε καθοριστικό ρόλο στη μεταρρύθμιση του ενίου χειριδίου κανόνων για τι ευρωπαϊκέ χρηματαγορέ και για την απόκριση στην ε, χρηματοπιστωτική κρίση, έσμα πιστεύω. Με τη δημιουργία αυτού του ενίου χειριδίου δημιουργήθηκε μια σειρά από δραστηριότητε εργαλεία και φορεί που από το 2011 μπόρεσαν να δώσουν 120 τουλάχιστον τεχνικά πρότυπα και 90 ε, σημεία τεχνικών συμβουλών με την επίβλεψη των, ε, ε, των οίκων ε, πιστοληπτικής αξιολόγησης μπορέσαμε να καθορίσουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης διαφάνειας και εσωτερικών ελέγχων με τις δύο περιπτώσεις τουλάχιστον σωστής επιβολής. Επίσης, οι εκθέσεις μας για τα παράγωγα και η επίβλεψη των κεντρικών αντισυμβαλωμένων από την, ε, από την ΕΣΜΑ ε, έδωσε πολύ, ένα διαφορετικό ε, πρίσμα για την αγορά παραγόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάλυψε και θέματα ποιότητας των δεδομένων. Το ίδιο και στην ατζέντα για την σύγκληση των εποπτικών αρχών των κατανομελών και τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε διαφορετικά εργαλεία, τρεις γραμμές, γνώμες, απαντήσεις και εκθέσεις ομοτήμων. Πιστεύω ότι έχουν ένα καλό συντονισμό στην περίπτωση αντιμετώπιση κρίσεων με μια ε, γρήγορη διαδικασία για να ε, ξεπεράσουμε τις ελλείψεις ε, τις εμπορικές συναλλαγές. Η ΕΣΜΑ ε, έχει βελτιώσει σημαντικά και την αντιμετώπιση των κινδύνων καθώς και τον εντοπισμό τους για την προστασία των επενδυτών. Έχουμε διαρκώς ε, βελτίωση στην συλλογή δεδομένων και θα ήθελα να σας ε, αναφέρω τώρα τα βασικά σημεία της θετικής μας για τα επόμενα χρόνια. Θα περάσουμε από την νομοθέτηση στην εφαρμογή πλέον. Η ΕΣΜΑ θα αφιερώσει περισσότερου πόρου στι διαδικασίε σύγκληση των εποπτικών αρχών και στι δραστηριότητε του ενίου εγχειριδίου κανόνων. Υπάρχει ε, περισσότερο περιθώριο για την σύγκληση των εποπτικών πρακτικών και προσεγγίσεων μεταξύ των εθνικών αριθμιστών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο στόχο μα είναι να έχουμε μια προσέγγιση που θα πρέπει ε, απαράλλακτη να εφαρμόζεται σε όλου. Θα πρέπει να δούμε την ε, σωστή εφαρμογή των ίδιων κανόνων και το κατά παρόμοιε παρόμοιες προσεγγίσεις, ε, παρόμοιε κινδύνου ωφελούν. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε για να επιτύχουμε του στόχου εγγύηση. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν προ διαφορετικού στόχου, όπω την αποτελεσματική υλοποίηση των κανόνων, την διευκόλυνση τη ανταλλαγή εμποριών μεταξύ εθνικών ε, ρυθμιστών, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων εποπτεία και την αποτίμηση των πρακτικών που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. το έργο σύγκληση τη εποπτεία θα είναι σημαντικό στοιχείο για την οικοδόμηση της, ε, της αγοράς κεφαλαίων της ε, Ένωσης Χρηματαγορών στην Ευρώπη με το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων επίση. Αυτό θα απαιτήσει ε, ένα μικρό μέρος των πόρων μας, αλλά θα, δώσει, θα αποτελέσει μια τεράστια πηγή εμπειρογνωμοσύνης για τις αγορές αξιογράφων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχετική νομοθεσία. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε τα τεχνικά πρότυπα του παρελθόντο και να τα προσαρμόσουμε όπου χρειάζεται στι νέε ανάγκε. Η συμβουλευτική και η επικοινωνία θα συνεχίσουν να είναι σημαντικέ για το έργο τη ΕΣΜΑ και στο ρόλο μου ω Προέδρου θα φροντίσω όλοι οι διάβλοι που υπάρχουν να αξιοποιηθούν μέσω τη ε, ομάδα των ε, ε, ενδιαφερομένων για, τις, για τα αξιόγραφα και τι αγορέ, με τι ανοιχτέ κροάσει, με τι διαβουλεύσει με το κοινό και συναντήσει με ενώσει από όλο το φάσμα δραστηριοτήτων με του ενδιαφερομένου από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε να επισκεπτόμαστε κράτη-μέλη για να έχουμε συζήτηση με του επενδυτέ, του φορεί τη αγορά και του εθνικού ρυθμιστέ. Για να πετύχουμε του στόχου σύγκληση, η ΕΣΜΑ θα ενισχύσει την ρυθμιστική συνεργασία σε επίπεδο ευρωπαϊκό και διεθνέ και γι' αυτό στηρίζουμε πλήρω και την αμυκτή Επιτροπή των ESA για, την, ε, για να εξασφαλίσουμε την εποπτική σύγκληση μεταξύ των τριών τομέων να υπογραμμίσω ότι η καλή συνεργασία της Επιτροπής σας με την ΕΣΜΑ θα συνεχίσει να είναι ζωτική σημασία. Θέλω να υπάρχει άτυπη ανταλλαγή απόψεων και, να, και μια μορφή συνεργασίας διαφανής και ανοιχτόμυαλη, όπως και ο ιδιωτικός μας κανονισμός προβλέπει. Θα πρέπει ε, μαζί να βεβαιωθούμε ότι η υλοποίηση της νομοθεσίας συνάδει με τους στόχους των συνομοθετών και συμβάλλει στους βασικούς στόχους οικονομικής ανάπτυξης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, συνεργασία που είχαμε τώρα. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας στο κοινό Κοινοβουλίο, ο κ. Ευχαριστώ. Κύριε Μάιο, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Κύριε Μαγιόρ, συχνά τονίζετε ότι μόνο ή περισσότερο ειδικό είσαι, τεχνοκράτης και όχι πολιτικός. Λέτε ότι εμείς είμαστε οι πολιτικοί θεσμοί. Η Κομισιόν είναι σημαντικό ότι πρέπει να είναι υπόλογη για μας για, την, για τις της πράξεις. Όπως και η ΕΖΑ είναι υπεύθυνη για να λογοδοτήσει σε εμάς για τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι φορείς εποπτείας λένε ότι υπάρχει περιθώριο ερμηνείας για αυτά που κάνουν και ότι δεν μπορούν να τα αποφασίζουν όλα μόνοι, μόνες τους, μόνοι τους αυτοί οι φορείς. Αναφέρονται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Διότι ξέρετε ότι πολύ συχνά συναντούμε αυτούς τους φορείς εποπτείας, όπως και το Συμβούλιο του συναντά. Οπότε η ερώτησή μου, πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι εποπτικοί φορείς ε, ε, βλέπετε να εξελίσσονται προς τεχνοκρατική κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Οι εποπτικοί φορείς είναι τεχνοκράτες, τεχνοκρατικοί φορείς ή πολιτικοποιημένοι. Εμείς είμαστε τεχνοκράτες ή πολιτικοί. Αυτά αναφέρονται στους ιδρυτικούς μας κανονισμούς. Οι εποπτικοί φορείς δημιουργήθηκαν για να είναι ανεξάρτητοι, να υπάρχει λοιπόν ανεξαρτησία στον καθορισμό των κανόνων και επίσης για να δώσουν και τεχνικές συμβουλές. Οπότε η εργασία μας είναι στην ουσία τεχνικής φύσης. Και αν δείτε πώς καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές στους ιδρυτικούς μας κανονισμούς, είναι τεχνική η φύση τους. Δεν είναι στρατηγική φύση. Προσπαθούν να αποπολιτικοποιήσουν το καθορισμό των προδιαγραφών. Αλλά τα τελευταία χρόνια, αν είμαστε ειλικρινεί, πρέπει να πούμε ότι μερικέ από τι αποφάσει που λήφθηκαν και κάποιε τεχνικέ προδιαγραφέ στην ουσία ήταν ε, ποιο θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι λοιπόν ε, έχουν κάπως διεισδύσει και κάποια πολιτικά στοιχεία στις τεχνικές μας ε, αποφάσεις. Επιμένω, εμείς είμαστε τεχνοκράτες. Πρέπει να έχουμε φυσικά πλήρη γνώση και συνείδηση των πολιτικών στόχων της πρωτογενούς νομοθεσίας. Δεν είμαστε καλοί πολιτικοί, εμείς μόνο καλοί τεχνοκράτες μπορούμε να είμαστε και το προσωπικό μας είναι τεχνοκράτες, ειδικοί. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά που αποφασίζουμε πρέπει να συμβάλλουν στο ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα πολιτικά στοιχεία της εργασίας μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντώτης. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια, για τη δουλειά σας, για τη δουλειά του προσωπικού σας και για τις αγωγικές σας τοποθετήσεις σε δύο τομείς. Θα ήθελα να αναπτύξω τις ερωτήσεις μου για το SM2 και το σύστημα Σύμφωνη 2. Η ΕΣΜΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξάφνιασαν την διαπραγματευτική ομάδα της ΕΚΟΝ ανακοινώνοντας ε, πως θεωρείται ότι θέλετε να αναβληθεί, ότι είναι καλύτερο να αναβληθεί η νομοθεσία για ένα χρόνο τουλάχιστον. Και αμέσω άρχισαν τα μέσα να ανακοινώνουν σαν να είχε ληφθεί η απόφαση αυτή την αναβολή. Δεν είναι σωστό αυτό και δεν νομίζω ότι είναι και ο σωστός τρόπος για να λαμβάνονται αποφάσεις τέτοιου τύπου με την ανακοίνωση αυτής του νομοθέτες. Έχω λοιπόν τα εξή ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ανακοίνωσε, γιατί δεν ανακοίνωσε νωρίτερα η ΕΣΜΑ. Είχαμε τόσες συναντήσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους αυτή την πρόταση για αναβολή στο Κοινοβούλιο, αφού ε, πέρασε και η προθεσμία της 3ης Ιουλίου για τη διαβίβαση των δεδομένων στην Επιτροπή, θα έπρεπε οπωσδήποτε να το πράξει. Επίσης πριν από έξι εβδομάδες εκφράσατε ανησυχίες για την εφαρμογή των ε, κανόνων του επίπεδου 2. Αλλά εγώ ενημερώθηκα γι' αυτό, επειδή κάποιοι από τα λόμπι του κλάδου είχαν λάβει από διαρροή αντίγραφα αυτών των προτάσεών σας και έτσι φτάσαν μέχρι εμένα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει απευθείας επικοινωνία. Και, βάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να έχουμε μια κατάσταση όπου η ΕΣΜΑ και η Επιτροπή προξενούν με δημόσιες ανακοινώσεις τέτοιες ε, εκπλήξεις σε επιτροπή και σε κοινοβούλιο και κοινοβουλευτική επιτροπή ενώ ο κλάδος είναι ενημέρος ακόμη και πιο νωρίς από εμά. Η κυρία Φερέρα επίσης ε, έχει εκφράσει κάποιες θέσεις για μια πλατφόρμα που θα επέτρεπε τη μόνιμη διαγραφή μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί ε, μεταξύ των παραγόντων της αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ για την... Με πρόεδρε αφήστε με τελειώσω, δεν έχω τελειώσει. Όχι, δεν γίνεται, λέει ο πρόεδρο. Ένα λεπτό έπρεπε να έχετε για τι ερωτήσει σα. Υπάρχουν και άλλοι και εσεί ξεπεράσετε τα δύο. Κυρία Ντότ, χωρί μικρόφωνο. Well, maybe start with the... Ας ξεκινήσω με την τελευταία σας ερώτηση το ζήτημα του σύμφωνη αυτής της πλατφόρμας. Για να απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Κεντρικό ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό υποχρέωση για διατήρηση δεδομένων συναλλαγών πληροφοριών, συνομιλιών και αυτά όλα περιγράφονται στην επιστολή. Μια πρώτη αντίδραση είναι η εξή. ότι προφανώς υπάρχουν υποχρεώσεις για διατήρηση ε, μητρώων αρχείων σχετικών με την επικοινωνία αυτή. Δεν παραβαίνουμε περισσότερο, αλλά προς το παρόν δηλώνουμε ότι φρονούμε πως υπάρχει μια σαφής νομική βάση και συνεχίζουμε με τους εθνικούς εποπτικούς φορείς τη συζήτηση, γιατί εκείνοι βεβαίως μπορούν να ε, επιτηρούν και την υλοποίηση. Θα δούμε αν υπάρχουν επιπλέον προβλήματα. Για την ε, διατήρηση αρχείων βεβαίως υπάρχουν πρακτικά ζητήματα αλλά εμείς πάνω απ' όλα θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε μια ισχυρή νομική βάση για τη διακράτηση αρχείων. Βεβαίως πρέπει το κομμάτι που θα έχει να κάνει με την εποπτεία αυτής της διακράτησης να παληθευθεί πιο συγκεκριμένα για το MIFID, για την ε, οδηγία MIFID και τις καθυστερήσεις. Αντιλαμβάνομαι βέβαια τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου εμείς και από το Διοικητικό του Συμβουλίου της ΕΣΜΑ ως συλλογικό όργανο, αλλά και εγώ προσωπικώς, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, ε, συνέπειες δυσάρεστες για μας και το Συμβούλιο, όπως έλεγα, και για μένα προσωπικά, από την καθυστέρηση αυτή την πρόοδο της νομοθεσίας. Το βλέπετε άλλωστε και από την επιστολή μας με την οποία επιχειρηματολογούσαμε υπέρ μιας πολύ στοχευμένης και συγκεκριμένη αναβολής μόνο για τα συστήματα πληροφορικής και όχι μιας πιο γενικής αναβολής. Γιατί το κάναμε αυτό. Διότι δεν θέλαμε να εγερθεί το θέμα στο δημόσιο διάλογο χωρίς να έχουμε σαφή εικόνα για το αν Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει το δικαίωμα της πρωτοβουλίας για τις αλλαγές θεωρούσε ότι είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν άρχισε η εποπτική αρχή, η ρυθμιστική αρχή να λέει Α, πρέπει να καθυστερήσουμε το συγκεκριμένο σημείο, αλλά δεν έχει το δικαίωμα τη πρωτοβουλία και εκείνη που έχει το δικαίωμα τη πρωτοβουλία, η Επιτροπή δηλαδή δεν συμφωνούσε, θα βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Ε, Πάντω αυτό προσπαθήσαμε να πούμε και βεβαίω σημειώνουμε ότι αν υπάρχει η πρόθεση, τότε πρέπει η ταχύτατα να εμπλακούν και οι συνομοθέτε στη δικασία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πω τι ευαισθησίε σα, αλλά και για να ολοκληρώσω, γιατί δεν ήταν δυνατόν να γίνει αξιολόγηση σε πιο πρώιμο στάδιο εδώ το συγκεκριμένο σημείο βασιζόταν στο ότι έπρεπε να γίνουν οι τεχνικές αξιολογήσεις μέχρι τελικού σταδίου. Συγκεκριμένα θα επιλέγαμε την EBA, την κόφια, αυτό συγκεκριμένα θα επηρέαζε τον κίνδυνο, της προδιαγραφές πληροφορικής και όλες τις λοιπές αποφάσεις που στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθούν. Στη λυπή διαδικασία, στη διαδικασία που θα ακολουθήσει δηλαδή. Αυτό τους δύο τελευταίους δύο με τρεις μήνες προχώρησε με τον εντοπισμό των αναγκών σε πληροφορική κάλυψη, σε δεδομένα και άλλαξαν τα στοιχεία άλλαξα ε, η περιγραφή των αναγκών τελευταία στιγμή, πρέπει να το πω αυτό ξεκάθαρα, και βέβαια υπήρξε και η πολιτική αξιολόγηση. Υπάρχει και η πολιτική αξιολόγηση ότι ίσως να μην έγινε η αποδοχή αυτών των προτάσεων το ταχύτερο δυνατό. Η κυρία Γουινμπέρν, ε, προφανώς ε, θα αντιληφθείτε ότι και εγώ θα συνεχίσω σχέση με τα προηγούμενα ερωτήματα. Ε, βλέπουμε να έχετε ε, κυρίως περιοριστεί στην έκδοση τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων του επίπεδου 2. Βέβαια υπάρχει ένα, μια πολιτική διελκυστίνδα στην υπόθεση αυτή ίσως έχει ασκηθεί από τα μέλη του Διοικητικού σας Συμβουλίου ε, και των Εθνικών Εποπτικών Αρχών να έχουν ληφθεί φάσεις και επιλογές οι οποίες ξεπερνούν τα όρια και πρέπει να επαληθεύεται, ε, πιστεύω, ε, το κατά πόσον τηρούνται οι προδιαγραφές κυρίως του επίπεδου 1 από το Διοικητικό Συμβουλίο και τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές. Μιλήσατε για τις ε, ερωταπαντήσεις, τις κατευθυντήριες γραμμές, ε, την τυποποίηση στα δεδομένα που θα επιτρέψει την γενικότερη εποπτεία της κατάστασης αγορές, τους συστημικούς κινδύνους κυρίως που μπορεί να εντοπίζονται αυτοί. Ερωτώ λοιπόν τι είδου εστίαση θα έχετε στις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές και ερωταποκρίσεις. Απάντηση. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, αλλά ξέχασα την πρώτη σας ερώτηση. Κύριε Σουίνμπερν. Ότι υπήρξαν ε, πολιτικές επιλογές. Τι θα πράξει σχέση με αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Για τα πρώτα στοιχεία. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό η δουλειά σε επίπεδο 2 να είναι συνεπής με τις επιλογές του επίπεδου 1. Το είπα κάπως χαριεντιζόμενος ότι θα έπρεπε να έχω έναν λογιστή ε, στο γραφείο μου που να μετράει κάθε μέρα τι λέμε και ε, τη συνέπεια με τα κείμενα του επίπεδου 1. Επομένως, σε σχέση με, το, με τη συνέπεια επίπεδο 2, επίπεδο 1, είναι μία εποδός την οποία ποτέ δεν λησμονούμε και πάντα επαληθεύουμε. Βεβαίως όμως πρέπει να αποδεχθούμε ότι είναι και ασαφή τα κείμενα, μερικές φορές δεν είναι ξεκάθαρο τι προθέσεις υπάρχουν στα κείμενα του επίπεδου 1 και επίσης ε, νωρίτερα ε, επισημάναμε ότι ήταν καλό να είχαμε παραπάνω πληροφορίες για τις ε, συνομιλίες στο τριμερή διάλογο, όχι γιατί είμαστε ε, μέρος των διαπραγματεύσεων, γιατί θα μπορούσαμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι σημαίνουν οι διατάξεις του επίπεδου 1. Και βεβαίως υπάρχουν αξιολογήσεις και νομικές προτάσεις του προσωπικού της ΕΣΜΑ, που αποτελούν νομική ερμηνεία. Και βεβαίω πολλές φορές έχουμε διαφωνήσει, έχει διαφωνήσει μάλλον η πλειονοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτό όταν θεωρήσαμε ότι δεν υπήρξε συνοχή και συνέπεια με το επίπεδο 1, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε μια διαφορετική ερμηνεία. Για το επίπεδο 1 λοιπόν αυτό. Για τις ερωταποκρίσεις Επιτρέψτε μου να πω το εξή, γιατί είχε τεθεί και νωρίτερα. Οι κατευθυντήριε γραμμέ και, και ερωταποκρίσει δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε ένα επιπλέον νομοθετικό ε, επίπεδο. Πρέπει να, πρέπει να υπάρχουν, γιατί μπορούν να επιτρέψουν την καλύτερη εφαρμογή τη νομοθεσία επίπεδου 1. Ε, αυτό όμω θέλω να επαναλάβω είναι ότι ε, η δουλειά μα είναι να εξασφαλίζουμε την συνέπεια με το επίπεδο 1 και η Επιτροπή βεβαίω τις ζητήσεις και με όσα ορίζει η συνθήκη οφείλουν, οφείλει να επαληθεύει, όπως και το Διοικητικό μου Συμβούλιο, τη συνέπεια, αλλά πρέπει να έχουμε και ταχαία συγκεκριμένα μέτρα που θα παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά και άρα χρειάζονται αυτές οι προτάσεις και οι ερωταποκρίσεις ως μέτρα σύγκλησης, ως εργαλεία. Φυσικά μπορούμε να επανέλθουμε και να συζητήσουμε μαζί σας όταν τα εκδίδουμε αυτά τα κείμενα και τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για να μας πείτε κι εσείς αν συμφωνείτε ότι εξασφαλίζουν τη συνέπεια. Και βέβαια η συλλογή δεδομένων και η μορφή με την οποία θα προσφέρονται θα είναι πολύ σημαντική και εκεί θα χρειαστεί να έχουμε μία συγκλίνουσα εφαρμογή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόρα Φανίδων Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ στην Επιτροπή, ε, σας καλωσορίζουμε εδώ στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και ως σχεδόν συγκήτρια για την, για την οδηγία 2 Πρέπει να πω ότι έχετε κάνει ήδη πολύ καλή δουλειά για ένα πολύ τεχνικό θέμα, για τη συγκριτική αξιολόγηση και τους δείκτες που χρησιμοποιούνται. Θα ήθελα λοιπόν να γίνουν πολύ περισσότερα ε, ε, και η ίδια προσπάθεια και για, τη, για τα διάφορα πρότυπα, όπως έχει γίνει για τους δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης. Στο θέμα των, ε, της επικοινωνίας τώρα που αναφέρατε και εσείς και στην ε, εκπόνηση τεχνικών προτύπων θέλουμε να πετύχουμε όλους τους στόχους εδώ χωρίς ε, πολιτική ανάμειξη. Οπότε η ερώτησή μου είναι θα βοηθούσε να γίνεται αυτή η συζήτηση κάπως πιο ε, εγκαίρος όταν τα προβλήματα αυτά αναδύονται σε πρώτη στη φάση προτού ε, ήδη δημιουργηθούν καταστάσεις και πρέπει να και καλείστε να απαντήσετε. Θα πρέπει λοιπόν ίσως να κινηθούμε εγκαίρος Ε, λόγου χάρη ε, κόφεα σε σχέση με το άλλο εργαλείο και με την λογοδοσία. Επίσης, στο επίπεδο 1 και τους σχετικούς κανόνες, ξέρουμε ότι εκεί είχατε μεγάλη συμμετοχή. Το ίδιο και για τις προτεραιότητες καλύτερης νομοθεσίας του κυρίου Τίμερμανς. Εκεί θα ήταν καλύτερο να υπάρχει η δική μας συμμετοχή ε, εγκαίρως. Σας ευχαριστώ. Θα απαντήσω και εγώ στα Ολλανδικά λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο σημείο. Πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε καλύτερη συμμετοχή στις συζητήσεις του επίπεδου 1. Το αναφέραμε επανειλημμένως ε, στους συνομοθέτες. Θέλουμε τέτοια συμμετοχή και, και περισσότερες διαπραγματεύσεις λαμβάνοντας ε, μέρος εγκαίρως της ε, συζητήσεις. Έχουμε συμμετάσχει σε συνεδρία στο Συμβούλιο στις Βρυξέλλες αλλά δυστυχώ χρειάστηκε να φύγουμε από την αίθουσα κάποια στιγμή όταν οι συζητήσει έγιναν απόρριτε. Τώρα για τη συνέπεια των κανόνων επίπεδου 1 και 2. Το έχω ήδη αναφέρει. Το να γίνονται σεβαστοί κανόνε στο επίπεδο 1 είναι ουσιαστική σημασία. Στι συζητήσει μα τον προηγούμενο μήνα τα συζητήσαμε εντελεχώ αυτά και του επίπεδου 2 και άλλα σημαντικά. Το ΣΧΕ. Που μπορεί να αποδειχθούν ευαίσθητα. Ίσως και αναδρομικά. Μπορεί εκ των υστέρων να καταλάβουμε ότι κάποιες νόρμες είναι ε, ίσως ακατάλληλες Εάν δούμε δηλαδή ε, τι γίνεται με τη MIFID, από τις 120 περίπου, 12 θα πρέπει να τις ξανασυζητήσουμε και ίσως ε, θα ήταν ε, καλύτερο να τις έχουμε συζητήσει εγκαίρως, όπως οι διαφάνειες προς τις υποχρεώσεις. Η υποβολή εκθέσεων για τα παράγωγα. όλα αυτά καλύτερα να είχαν προλευθεί εγκαίρως. Ευχαριστώ. Ο Σβέν Γκίγκολτ. Καλώ ήρθατε και από πλευρά της ομάδας μου. Σε δύο θέματα θα αναφερθώ. Θεωρείτε ότι θα, μπορούσαν να υπάρ... θα να υπάρξουν κοινέ προσπάθειες υποβολής εκθέσεων από τους τρεις εποπτικούς οργανισμούς για την επιλογή δικαιοδοσίας. Και να επανέλθω σε αυτά που είπε Ανελίζε για τα προβλήματα που έχουμε με το MIFID. Θεωρείτε ότι είναι ακόμη καλή ιδέα να βάλουμε σε μία δέσμη τις διάφορες προδιαγραφές. Άρα, γιατί αυτό, ξέρετε, μπορεί να δώσει δυνατότητα διακανονισμών που δεν ήταν στις, στις προθέσεις των νομοθετών. Και δεύτερον, πώς θα ανταποκριθείτε πώς θα αντιμετωπίσετε τις διαρροές είτε από το δικό σας θεσμικό όργανο είτε από άλλους θεσμούς μπορείτε να δεσμευτείτε ότι και εσείς και το προσωπικό σας θα αναφέρουν όλες τις επαφές που έχουν με τον κλάδο διότι ξέρετε ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση να υπάρχει λιγότερη διαφάνεια στους δικούς οργανισμούς από ό,τι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις επαφές με τα λόμπι. Απάντηση. Για τον σκιώδη τραπεζικό τομέα. Δεσμεύομαι μαζί με τον Γκάμπριελ και τον Ανδρέα να σας δώσουμε μια επισκόπηση του τι έχουμε κάνει για τον τομέα αυτό. Γιατί είναι σημαντικό να αντιληφθείτε ότι ήδη έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα και από διάφορες ε, οπτικές γωνίες. Και εμείς και τα άλλα εποπτικά όργανα ασχολούνται πολύ με διάφορα θέματα του τομέα αυτού και στον Οργανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στον ΙΟΣΚΟ πρέπει να καταλάβετε ότι πολλές μεταφορές κεφαλαίων σε όλα τα τμήματα και από όλα τα τμήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα οφείλονται κυρίως στα χαμηλά επιτόκια. Άρα ένα μεγάλο τμήμα αυτών που φεύγουν από τον τραπεζικό τομέα και πηγαίνουν στο μη τραπεζικό τομέα έχουν να κάνουν με τα χαμηλά επιτόκια και τη δουλειά που έχει γίνει από τα θεσμικά όργανα ένα μεγάλο τμήμα του μη τραπεζικού τομέα είναι ήδη υπό επιτήρηση βέβαια σε αρχική φάση πάντα έχουμε εξετάσει και τα εναλλακτικά ταμεία βέβαια δεν έχουμε ολοκληρώσει την ε, εξέτασή μας βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε και τις δοσοληψίες ε, ρήπο και το δανεισμό αξιογράφων. Ένα μεγάλο τμήμα λοιπόν του μη τραπεζικού τομέα είναι ήδη υπό εποπτεία και ήδη υπάγεται σε κανονιστικές διατάξεις. Αυτό δεν αφορά αυστηρά τον ε, σκιώδη τραπεζικό τομέα. Έχει να κάνει και με την επιλογή δικαιοδοσίας, εποπτικής. Και από πλευρά των καταναλωτών πρέπει να το δούμε αυτό. Πιστεύω ότι και ο ασφαλιστικός τομέας πρέπει να έχει τις ίδιες πρακτικές πωλήσεων όπως ο τομέας των κινητών τίτλων. Δεν έχουμε διασφαλίσει ομοιόμορφους κανόνες. Τώρα για τις διαρροές. Είμαι απόλυτα σαφής. Με δυσαρεστούν ιδιαίτερα αυτές οι διαρροές. Παραβαίνουν τους κανόνες μας, τις δεσμεύσεις μας που αναφέρονται και στον ιστοτόπο μας όπου όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύονται να τηρούν την εμπιστευτικότητα. Εάν δεν το λύσουμε αυτό, δεν θα είναι βιώσιμη η περαιτέρω λειτουργία μας. Πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γιατί θα έχουμε περισσότερα προβλήματα. Όπως είπατε, οι διάφορε επιχειρήσεις του κλάδου ξέρουν τι γίνεται και το κοινοβούλιο δεν το ξέρει. Πρέπει να το λύσουμε αυτό. Το καταλαβαίνω πλήρω. Ότι δεν είναι βιώσιμη η συνέχιση αυτή της κατάστασης. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει νωρίτερα ο κλάδος έγγραφα από ότι εσείς. Βεβαίω, θα συζητήσουμε με το προσωπικό μας, θα συζητήσουμε με τις επιχειρήσεις με τις οποίες είμαστε σε επαφή, και θα γνωστοποιήσουμε την αντίδραση του κάθε οργανισμού με τον οποίο είμαστε σε επαφή για να υπάρξει σαφήνεια. Όπως είπε και ο εκτελεστικός διευθυντής που εκπροσωπεί το προσωπικό, αλλά και εγώ θέλουμε να είμαστε πλήρως διαφανείς στις επαφές που έχουμε με τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ευχαριστώ, Νταϊάν Καλημέρα και ευχαριστώ που ήρθατε. Την προηγούμενη εβδομάδα ρώτησα τον κύριο Ντράγκη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εάν διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας δεν ήταν διτεθειμένος να έρθει σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή, αν ε, κρυθεί αυτό απαραίτητο για να εξηγήσει την κατάσταση. Ισχυρίστηκε ότι δεν αντελήφθη την ερώτησή μου. Αυτό θεώρησε καλύτερο. Ένας από τους ε, επικεφαλής άλλης ρυθμιστικής ε, αρχή, της ΕΤΑ, Μα είπε σήμερα ότι βεβαίω και θα ερχόταν. Εσεί λοιπόν μπορείτε να μα πείτε αν υπάρχει κάποιο λόγο να μην έρθετε ενώπιον Εθνική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να εξηγήσετε ε, ζητήματα που μπορεί να φέρουν το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμέτωπο ως προς την ε, ρυθμιστική του αρχή με αυτήν ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απάντησε. Έχω πάει ενώπιον επιτροπών εθνικών κοινοβουλίων πολλές φορές και και τι αναγνωρίζω ότι ε, έχω υποχρέωση λογοδοσίας μόνο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ε, καλές και τακτικές επαφές και με τα κράτη-μέλη, με τις αρχές τους, με τις μυστικές αρχές, με τα κοινοβούλια ενδεχομένω όπως συχνά ε, καλούμεθα να πράξουμε ανταλλαγές απόψεων, με κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, τα ισοδυναμά δηλαδή τη επιτροπή σα σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια όλα αυτά επιτοπλίστων επικεντρώνονται σε ζητήματα πολιτικής και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι δύσκολο να δώσω απάντηση σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μιας εξεταστικής επιτροπής. Το 70-80% της δουλειάς μας, ξέρετε, έχει να κάνει με ρυθμιστικά ζητήματα με προσδιορισμό δηλαδή κανόνων και μέχρι τώρα δεν έχουμε κληθεί σε εξεταστική επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος Μπερνάρ Μονό. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σα. Η ΕΣΜΑ έχει ήδη υπό τη διοίκησή σας αποτύχει την εντολή, στην εντολή που της έχει ανατεθεί, δηλαδή να ρυθμίσει την αγορά. Ήδη έχετε ξεκινήσει μία πρόταση, με καθυστέρηση βέβαια του ΕΜΙΡ, ε, για την αναθεώρηση της ε, ΜΥΦΙΤ, για να προετοιμάσετε υποτίθεται τις αγορές. Και φαντάζομαι ότι θα σας δοθεί αυτή, θα δοθεί αυτή η παράταση που θα επιτρέψει έως το 2018 να συνεχίσει το City του Λονδίνου τις ε, μη διαφανείς δραστηριότητες. Η ΕΣΜΑ βλέπουμε να καθυστερεί δίνοντας πλεονέκτημα στις αγορές του Λονδίνου και στους φορείς του Λονδίνου. Αυτό είναι σκάνδαλο και αν είμαστε στον ιδιωτικό τομέα με δεδομένα τα αποτελέσματα της δουλειά σας θα σας είχαμε ήδη απολύσει και γι' αυτό και η ομάδα μου δεν υποστηρίζει την ανανέωση της εντολής σας για την ΕΣΜΑ. Ευχαριστώ πολύ και επιτρέψτε μου πρώτα να υπογραμμίσω πως πιστεύω ότι και το προσωπικό της ΕΣΜΑ αλλά και το Διοικητικό μου Συμβούλιο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει εκδώσει τεχνικές προδιαγραφές και συμβουλές τα τελευταία χρόνια, εν πάνω από 200, 200 ε, έγγραφα τεχνικών προτεγραφών και συμβουλών, στην ώρα τους τα περισσότερα, με μια καθυστέρηση μόνο τριών μηνών σε σχέση με την πτυχή αγορά της ΜΕΦΙΤ, πράγμα το οποίο όμως σχετιζόταν και με την ανάγκη για μια πρόορη αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που χρειαζόταν να προχωρήσει και βέβαια πρέπει να συνεργαστούμε σε αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τρίμηνη αυτή καθυστέρηση έχει να κάνει με την αναθεώρηση των νομικών κειμένων, των νομοθετικών κειμένων. Ε, στην επιστολή δε που συστήθηκε νωρίτερα είχαμε ιδιαίτερα επισημάνει μια ανάγκη για περισσότερο χρονικό διάστημα προθεσμίες σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής για το καθεστώς διαφάνειας και για τις εκθέσεις διαφάνειας. Θα το δείτε και αργότερα αλλά στο κείμενό μας. Το έχω πει νωρίτερα και με τις συζητήσεις της ΜΥΦ. Ήταν καθαρά τεχνικά τα στοιχεία στα οποία εστιάζαμε το αίτημά μας και δεν είχαν να κάνουν με τη γενικότερη λογική της ΜΥΦΙΤ. Και επίσης ήθελα να πω ότι η πρόταση για καθυστέρηση ενός έτους που αναφέρετε εσείς είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ μακρύτερη από αυτή της τρίμηνης καθυστέρησης στην οποία αναφέρθηκα εγώ. Αυτό προκύπτει από τις συνομιλίες, από τον τρόπο με τον οποίο είχαν διατυπωθεί τα κείμενα, που οδήγησε στο συμπεράσμα ότι θα χρειαστεί περισσότερο από ένα χρόνο, μάλλον μια μακροχρόνια περίοδο, δηλαδή ένα χρόνο για να υλοποιηθούν οι ε, αλλαγέ αυτό γιατί, γιατί κινδυνεύαμε να έχουμε κακή εφαρμογή, προβληματική κατάσταση, απουσία συνοχή και συνέπειε σε αγορέ. Γιατί πρέπει και εμεί βέβαια να συλλέγουμε τα δεδομένα, αλλά εμεί ω εποπτικέ αρχέ, αλλά ε, και τα δεδομένα αυτά να είναι τέτοια που να επιτρέπουν και στι αγορέ να λειτουργούν. Γιατί διαφάνεια φερειπίν των τίτλων, η αγορά θα γνωρίζει μόνο ποιοι είναι αυτοί οι τίτλοι οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές διαφάνειας όταν έχουμε το, τη δυνατότητα να συλλέγουμε τα σχετικά στοιχεία. Ευχαριστώ κύριο Φαντέν Κελνάρε. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μα. Έχω μια ερώτηση για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο. Η ΕΣΜΑ ξέρουμε ότι κάνει πολλά για να επιτρέψει το Κοινοβούλιο να εκτελεί τον δημοκρατικό έλεγχο για τα μέτρα του επίπεδου 2. Αλλά δεν αρκούν. Αυτά πρέπει να γίνουν κι άλλα. Ο άλλο νομοθέτη φαίνεται να επηρεάζει από τη λένε ορισμένοι. Επίσης ε, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι λαμβάνει υπερβολικά υπόψη η ΕΣΜΑ της, ε, το, τον τραπεζικό κλάδο. Ε, και νομίζω, το χρηματοπιστωτικό καλύτερα κλάδο, και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστή ισορροπία δυνάμεων σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εσείς τι έχετε να μας πείτε, πώς μπορείτε να απαντήσετε στις επικρίσεις αυτές. Απάντηση. Κοιτάξτε, όπως είπε και ο Ανδρέα Ενρία, στη δική του παρέμβαση νωρίτερα σήμερα. Με ξεφνιάζει η εντύπωση που περιγράφεται ότι έχουμε πιο στενές σχέσεις με το Συμβούλιο από ότι με το Κοινοβούλιο. Διότι είναι σαφές και μάλιστα πάνω απ' όλα σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ δεν εμφανίστηκα ποτέ σε σύνοδο ολεμελίας του Συμβουλίου. Και αυτό άλλωστε προβλέπεται και από την ιδρυτική μας πράξη, από τον ιδρυτικό κανονισμό. Εγώ είμαι υποχρεωμένο να προσέρχομαι στο Κοινοβούλιο για να λογοδοτώ, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται για τη σχέση μου με το Συμβούλιο. Ε, επιτρέψτε μου λοιπόν να διαφωνήσω με την ε, ιδέα και τον υπενιγμό ότι μπορεί να έχουμε περισσότερες επαφές και συχνές ε, συνομιλίες με το Συμβούλιο. Ίσως μάλιστα αν δείτε μπορεί και εκείνοι να έχουν την ίδια εντύπωση. Γιατί τώρα τελευταία μου ζήτησα να πηγαίνω πιο συχνά στο Συμβούλιο βλέποντας ότι έχουμε αρκετά συχνέ επαφέ. Ε, με το Κοινοβούλιο φαίνεται πως επιδιώκουν και εκείνοι περισσότερη επικοινωνία. Όταν αρχίζετε εσείς, αρχίζουμε εμείς να συζητούμε περισσότερα θέματα της ΜΥΦΙΤ, βλέπουμε ότι προξενήσατε και μια αντίδραση από το Συμβούλιο που θέλει και εκείνο συχνότερες επαφές. Αυτά νομίζω ότι πάντα βέβαια με σεβασμό της ισορροπίας της επικοινωνίας και με μια πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, νομίζω ότι δεν υπάρχει εμβολία και δεν είμαστε πιο διαφανείς έναντι του Συμβουλίου από ότι έναντι του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Πέχμα σου πέχα τελευταία ερώτηση. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι. Είστε υποψήφιος για παράταση της εντολής και της θητείας. Για τις ε, κεφαλαϊκές αγορές και την κεφαλαϊκή ένωση δεν βλέπω να σχολιάζει κανείς την ε, ενίσχυση της ε, δύναμής τους και θα ρωτούσα τι έχετε να προτείνετε και επίσης για την προστασία των καταναλωτών γιατί πολλά ακόμα μένουν να κάνουμε Καθώς είμαι συγγήτρια για το σχετικό θέμα, θέλω να ρωτήσω το εξή, ε, γιατί θυμάμαι πολύ καλά και τις διαπραγματεύσεις που είχαμε μαζί με τους κοιόδης συγγητές για το ζήτημα των χρονικών αναφορών αξιολόγησης κινδύνου. Και δεν αποκλείστηκαν ποτέ οι ιστορικές αναφορές στις εργασίες μας. Τώρα όμως φαίνεται να έχουν απαλληφθεί οι παρελθούσες επιδόσεις και να έχουμε μόνο προβολές επιδόσεων στη νέα πρόταση. Αυτό θα ήταν ε, ε λάθος επιλογή και θα ε, μας εμπόδισε από το να βλέπουμε τις πραγματικές επιδόσεις και την ποιότητα των αγορών. Επίσης η αναφορά για τις ασφαλίσεις ζωής. Οι διατάξεις οποίες εμείς Στη νομοθεσία για την ε, νομοθεσία που κάλυπτε της ε, USIT, της OPSVM, είχαμε προτείνει υποχρέωση για τον εκδότη να περάσει στην πράξη σε ένα νέο σύστημα. Πώς μπορούσε δηλαδή να οργανωθεί η μετάβαση μεταξύ των δύο αυτών νομοθετικών ε, διατάξεων και βέβαια πάντα για την προστασία του επενδυτή, βλέπω με ανησυχία ένα, ένα προϊόν, το Forex, το οποίο πωλείται στον ιδιώτη. Ένα προϊόν λοιπόν με το οποίο υποτίθεται ότι θα γίνει trader μέσα σε μία μέρα ο ιδιώτης. Πωλείται πολύ στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, ακόμα και την Ισπανία το Forex. Ερωτώ λοιπόν τι είδους συντονισμό σκοπεύει να ε, προβλέψει ΕΣΜΑ για το θέμα αυτό, ποιες είναι οι εξουσίες που μπορείτε να ασκήσετε και μήπως δεν έχετε επαρκείς εξουσίες για να επιτελέσετε το έργο σας σε μια τέτοια περίπτωση. Ας ξεκινήσω με την τελευταία σας ερώτηση. Όντως βλέπουμε να να πουλούνται εξωτικά θα τα πω εγώ προϊόντα, όλη, με την ανετική έννοια βέβαια εξωτικά προϊόντα ε, έχουμε προϊόντα ε, συναλλάγματος, ε, διοικές επιλογές, binary options και πολλά άλλα. Το βλέπουμε όλο και περισσότερο επειδή σχετίζονται με τις διασυνοριακές προβλέψεις, διατάξεις για τον επενδυτή από τη χώρα της έδρας, πώληση σε χώρα υποδοχής. Αυτό που κάνουμε λοιπόν για αυτούς τους τομείς των προϊόντων είναι να καλούμε τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, κατά, χώρο, κατά, κατά τόπον αρμόδιες, για να εξετάσουμε την κατάσταση. Γιατί κάποιοι εκ των κινδύνων για, την, για παραβίαση των κανόνων της MIFID πραγματοποιούνται στη χώρα υποδοχής και άρα με αυτή τη ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί εκείνη θα είναι η αρχή η οποία εν τέλει θα πρέπει να επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. Άρα αυτό μπορώ να πω συνοπτικά είναι ότι έχουμε πολύ στενή συνεργασία. Φέρνουμε σε επαφή τις ρυθμιστικές αρχές έδρας, προελεύσεως και υποδοχής από κοινού. Παρακολουθούμε αυτές τις δραστηριότητε και ταυτόχρονα καλούμε τον... Δεν θα έπρεπε, λέει η κυρία Περές, να απαγορεύονται αυτά τα προϊόντα. Ναι, να σας πω το εξής. Ε, αυτός ο συντονισμός γίνεται σε εκούσια βάση Ταυτόχρονα σαφές είναι ότι αυτή η ίδια μεσολάβηση που έχει δεσμευτικό χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο οδηγεί τις εθνικές αρχές τις σωστές επιλογές. Η απαγόρευση θα έρθει με τον BFIT 2. Εκεί προβλέπεται η δυνατότητα απαγόρευσης. Χωρίς να λέω ότι αυτά τα προϊόντα θα επιλεγούν για απαγόρευση, αλλά πάντως θα έχουμε τη δυνατότητα να τα απαγορεύσουμε. Για την παρατήρηση σχετική με τις επιδόσεις. Ναι, βεβαίως αντιλαμβανόμεθα ότι οι ιστορικές επιδόσεις έχουν με την πρίψη λιγότερο, μικρότερο ρόλο από ότι με τη usage. Ωστόσο πρέπει και μια και έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά να πούμε ότι χρειάζεται να είναι σαφέστερη η νομοθεσία του επίπεδου 1 σε σχέση με τις ιστορικές πληροφορίες. Τώρα σε σχέση με το περιβάλλον usage. Ευχαριστούμε, οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτήν την ε, κρόαση. Σας ευχαριστούμε για την ανταλλαγή απόψεων και για αυτή την επικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή So we start now uh, our hearing uh, with uh, the executive directors. First is Adam Farkas, the EBA executive director. Και τώρα συνεχίζουμε τον κύριο Φάρκας, εκτελεστικό διευθυντή της EBA. Καλώς ήρθατε και σας καλώ να περιοριστείτε αυστηρά στα 5 λεπτά για τις αγωγικές σας παρατηρήσεις για να συνεχίσουμε μετά με ερωτήσεις και απαντήσει από ένα λεπτό η καθεμία. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, μέλη τη Επιτροπή, θέλω να σα ευχαριστώ που με προσκαλείτε στην Επιτροπή σα για να σα δώσω μια επισκόπηση των κύριων οργανωτικών επιτευγμάτων τη ΕΤΑ ω νέο ανεξάρτητο σώμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα θέλω να επικεντρωθώ στι δραστηριότητε για την επόμενη πενταετία. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τους περιορισμούς των πόρων που σημαίνουν σημαντικούς ε, Σημαντικέ προκλήσεις για τον εκτελεστικό διευθυντή. Έχουμε επιτύχει λοιπόν τη μετάβαση από τη CBS σε μια πλήρη ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνε και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στην αρχή μας ε, και, και έχουν θεσπιστεί τα όργανα, τα διοικητικά. Έχουμε πενταπλασιάσει τον οργανωτικό μα όγκο με πολύ σημαντική αξιοποίηση προσωπικού με διάφορους τύπους ε, συμβάσεων απασχόλησης, εργασίας καλύτερα και ε, με, ε, με τη διατήρηση υψηλής ποιότητας και κινήτρων προσωπικού έχουμε δημιουργήσει την υποδομή, αποτελεσματική υποδομή σε πληροφοριακά συστήματα και επικοινωνίες. Υποδομές επίσης που έχουν να κάνουν με την ε, παραγωγή εκθέσεων ε, ρυθμιστικών και προληπτικών, με την συλλογή των δεδομένων και τις αναλυτικές δυνατότητες που ε, μας χαρακτηρίζει. Ο προγραμματισμός και η διαχείριση ενός πολύ πυκνού προγράμματος εργασίας της ΕΒΑ έχουν, της έχουν ιδιαίτερα βελτιώσει, έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με την με το χρονισμό της παραγωγής ε, των προϊόντων που ορίζονται από την εντολή μας η διαφάνεια των διαδικασιών, οι πολιτικές επιλογές, το ενολυτικό έργο έχουν κερδίσει το σεβασμό όλων των εμπλεκομένων παραγόντων και έχουμε βεβαίως αντιμετωπίσει ως μεγαλύτερη πρόκληση το ζήτημα του προσωπικού παρά την ιδιαίτερη υποστήριξη από την Επιτύπωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί ουσιαστικό κίνδυνο για την υλοποίηση της εντολής μας και την διασφάλιση της αξιοπιστίας μας. Αυτό οφείλεται στην ε, προσήλωση του προσωπικού μας σε κάθε επίπεδο, που δημιουργεί έτσι ένα θετικό επαγγελματικό περιβάλλον παρά τις πιέσεις και το άγχος, ε, σε σχέση και με τις εθνικές αρχές, με βραχυπρόθεσμη υποστήριξη κατά κύριο λόγο σε συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής πέραν των επιτεύγματων σε σχέση με την τραπεζική νομοθεσία στην Ευρώπη και για να απαντήσουμε και στην οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση με την αναλυτική μας δουλειά και την συγκλητική και την εποπτική σύγκληση που επιδιώκουμε, έχουμε δραστηριοποίηση νέα μέσα, διαμεσολάβηση, διαδικασίες παραβίασης του δικαίου, έχουμε συλλέξει μια σειρά από προσφυγές και ε, παράπονα σε σχέση με το πεδίο αρμοδιοτήτων μας, αλλά έχουμε κάνει και διατομεακές παρεμβάσεις, επιτεύγματα τα οποία αναγνωρίστηκαν στην πρώτη γενική αναθεώρηση και επισκόπηση του έργου της CBA το 2014 από τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Τώρα για την επόμενη πενταετία θα ήθελα να πω ότι βέβαια η υλοποίηση του ρυθμιστικού, ε, των ρυθμιστικών εντολών και η ολοκλήρωση του εγχειριδίου, ε, του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων ε, έχει να ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά πρέπει να μετακινήσουμε το επίπεδο, του ονιστίαση των δραστηριοτήτων μας προς την παραγωγή ε, πιο τεχνικών και εις βάθος έργων για πιο σταθερή λειτουργία, πιο αποτελεσματική λειτουργία της τραπεζικής αγοράς και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν η έντα θα προχωρήσει με το ρυθμιστικό πλαίσιο, θα περιορίσει τη διακριτική ευχέρεια και το, τις αποκλήσεις της ερμηνείας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε έτσι την συνοχή στην εφαρμογή του εγχειριδίου κανόνων και να εξασφαλίσουμε τη μετακίνηση της απασχόλησης του εργατικού μας δυναμικού, στην απάντηση που θα πρέπει να δοθεί μετά την κρίση, στην περίοδο μετά την κρίση και βέβαια ταυτόχρονα την υλοποίηση του ε, θεσμικού πλαισίου στο οποίο στηρίζεται η ίδρυσή μας η σύγκληση, η ανάλογα η απουσία σύγκληση εποπτικές αρχές και οι συνέπειε αυτή στην ενιαία αγορά είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει. Θα έχουμε θεματική κατάρτιση, θα έχουμε επισκόπηση από τους ομότιμους, θα έχουμε επίσης αξιολόγηση κινδύνων και τακτική παραγωγή εργαλείων τεστ αντοχής Υπάρχουν εργαλεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος με υψηλή διασύνδεση με τον τραπεζικό τομέα. Επίσης, τα μέτρα για την προστασία του καταναλωτή, η χρηματοπιστωτική καινοτομία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, επιχειρησιακά πρότυπα ε, και η προτεραιότητα θα πρέπει να παραμείνει στην διαχείριση της τραπεζικής κρίσης, προγραμματισμό και διευκόλυνση δηλαδή της εκτέλεσης των μέτρων διαχείρισης της κρίσης εν όλο στην επόμενη πενταετία επαγγελματικά, τεχνικά και οργανωτικά αναμένουμε να έχουμε προκλήσεις εξίσου σημαντικές αλλά και ελκυστικές όπως και στην προηγούμενη, στην προηγούμενη περίοδο και ελπίζω ότι θα μπορέσω να συνεχίσω το έργο αυτό με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Κάρας. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτη. Θα ήθελα να μου πείτε για πόσες τράπεζες είναι αμφίβολο εάν τηρούν τους ε, κανονισμούς με βάση τους κανονισμούς μας και με βάση το Βασιλεία 3 και τι επιπτώσεις θα έχει για όσους δεν τηρούν τους κανόνες. Δεύτερον, αναφερθήκατε στα τεστ αντοχής του 2014 που έγιναν σε 120 τράπεζες και προτίθεστε το 2016 να ελέγξετε 153 τράπεζες. Συγγνώμη, είχατε κάνει πολύ περισσότερους ελέγχους στο 53... Α, θα μειωθούν σε 53 το 16 από τις 120. Γιατί μειώνεται τόσο πολύ. Θα ήθελα να μου πείτε επίσης τι ρόλο παίζει το χρέος τους προς ε, το, τα τμήματα του ενεργητικού τους που είναι κρατικά ομόλογα. Τι δουλειά έχει κάνει η ΕΜΠΑ για ένα πρότυπο για να ληφθεί υπόψη ακριβώς αυτός ο κίνδυνος από τα κρατικά ομόλογα. Thank you. Um, thank you Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, τις ερωτήσεις σας. Θα είμαι σύντομος. Για το κανονισμό για τα μπόνους, όπως ξέρετε, η EBA πρέπει να κάνει τακτικά εκθέσεις για τις αμοιβέ των ε, διοικητικών στελεχών και του προσωπικού των τραπεζών. Έχουμε αιτήσει τέτοιες εκθέσεις. Ξέρετε επίσης ότι είμαστε στη φάση αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραμμών για τις αμοιβέ για τον τραπεζικό τομέα και από αυτή την άποψη κάναμε μία έκθεση για την πρακτική των τραπεζών και μερικά από τα ευρήματα των εκθέσεων σαφώς καταδεικνύουν ότι υπάρχουν θέματα. Για παράδειγμα υπάρχουν διάφορα επιδόματα θέσεις σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν γίνονται με βάση διάφορα κριτήρια. Εάν λοιπόν δεν γίνονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τότε θεωρούμε ότι είναι μπόνους. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο ελέγχουμε τη συμμόρφωση προς αυτούς τους κανόνες είναι αρμοδιότητα των εποπτικών αρχών που επιτηρούν τα ιδρύματα και ε, βλέπουν τι συμβόλαια έχουν συνάψει με το προσωπικό τους. Για τα τεστ αντοχής, το δείγμα για το 2016 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την EBA όντως περιέχει μόνο 53 τράπεζες. Τα κριτήρια που χρησιμοποίησαμε μαζί με τις αρμόδιες αρχές συμπεριλαμβανομένου του SSM ήταν να καλύψουμε κατά 70% την τραπεζική αγορά και 70% των ε, εθνικών αγορών. Μία σημαντική εξέλιξη είναι το SSM αποφάσισε ότι βάση αναφοράς για την αγορά για να καλύψουμε δηλαδή το 70% θα είναι η Ευρωζώνη, όχι οι μεμονωμένες χώρες. Και κάτι άλλο είναι ότι για ορισμένες μικρότερες χώρες, όπου υπάρχει κυρίαρχη θέση των θυγατρικών κάποιων διεθνών τράπεζες, θα είναι κάπως χαμηλότερη κάλυψη, γιατί αυτές οι θυγατρικές θα ελεγχθούν σε ενοποιημένο επίπεδο, στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης της Ένωσης. Με βάση αυτά τα κριτήρια και μερικά συντροματικά, που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση τραπεζών, ή κάποιες μεμονωμένες τράπεζες που θεωρούνται ότι έχουν συστημικό χαρακτήρα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν με βάση όλα αυτά μειώσαμε σε 53 τις τράπεζες το δείγμα. Θεωρούμε με τη Συμφωνία για των Αρμοδίων Αρχών ότι ελέγχοντας αυτές τις αρχές ε, ελέγχουμε πολύ σωστά και αντιπροσωπευτικά το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα μέσω αυτών των επερχομένων ε, ελέγχων για τον κίνδυνο έκθεση στο, στα κρατικά ομόλογα. Από προληπτική πλευρά η δημιουργία, η έκδοση των ομολόγων ελέγχεται από διάφορες ε, πλευρές και παγκοσμίως και στην Ευρώπη και είναι απόλυτα σαφές ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί το πώς αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος από τα κρατικά ομόλογα. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό από προληπτική άποψη. Αυτή τη στιγμή επανεξετάζεται αυτό το πλαίσιο στη Βασιλεία αλλά και στην Ευρώπη. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου που εξετάζει ακριβώς αυτό το θέμα. Και επιπλέον υπάρχουν και εθνικές αξιολογήσεις και διάφορες προτάσεις σε εθνικό επίπεδο. Αλλά αυτή η εργασία δεν έχει καταλήξει ακόμη και δεν υπάρχει συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή πρόταση για αλλαγές του ε, ισχύοντος πλαισίου στην Ευρώπη. Ευχαριστώ η Ελίσσα Φερέιρα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα πώς διαχειρίζεστε τις σχέσεις σας με τον SSM και τον SRM. ιδιαίτερα ε, στο εγγύς μέλλον όταν μετά την 1η Ιανουαρίου θα έχουμε τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης έχουμε τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας και μετά την εφαρμογή των κανόνων διάσωσης με συμμετοχή των καταθετών κάποιες τράπεζες θα πάνε στα χέρια του μηχανισμού εξυγίανσης και ένα μεγάλο στοιχείο των κεφαλαίων τους θα είναι κρατικά ομόλογα. Θα έχουμε λοιπόν ε, μία αλλαγή στην κατάσταση. Πώς λοιπόν προβλέπετε να αντιμετωπίσετε τα χαρακτηριστικά κινδύνου και τι συστάσεις θα υπάρξουν σε σχέση με αυτές τις τράπεζες. Μία δεύτερη ερώτηση. Πάλι σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα. Αν ζητηθεί, ας πούμε, οι τράπεζες να μειώσουν την έκθεσή τους σε κρατικά ομόλογα, σε κρατικό χρέος. Και αν χρειαστεί να υπάρξει ε, μαζική πώληση ομολόγων, τι επιπτώσεις θα έχει στην αγορά. Πώς θα επηρεαστεί η συστημική βιωσιμότητα του τομέα αυτού, γιατί αυτό είναι ένα συνολικό θέμα. Θα έχει μακροοικονομικές επιπτώσεις. Το έχετε εξετάσει καθόλου. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ τα ερωτήματα αυτά θα μπορούσαμε να συζητάμε ένα ολόκληρο πρωινό. Είναι πολύ ευρέως φάσματος για SSM και SRM. Να σας πω κάτι, μια ιστορία. Φυσικά υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας μεταξύ αυτών των οργανισμών και ημών. Αλλά γενικά η Τραπεζική Ένωση, όπως είπε και ο Ανδρέα στη δική του ε, εισαγωγή, αλλάζει την κατάσταση η δημιουργία ενός ε, ενιαίου μηχανισμού εποπτείας και ενός ενιαίου μηχανισμού εξυγένσης θα προκαλέσει σοβαρή εμβάθυνση της ενοποίησης ε, την Ευρώπη παρά το ότι θα αφορά μόνο ένα περιορισμένο αριθμό κρατών, όχι όλες τις χώρες της Ένωσης. Πώς συνεργαζόμεθα με τον ε, SSM και τον SRB. σχέση που τους θέτει εντό του μηχανισμού ε, εποπτείας και εξυγίανση, συγγνώμη, εξυγίανση και ανάκαμψης, είναι το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων. Αυτή είναι η βάση για όλους τους αρμόδιους επιτηρητές. Ο SSM και η δημιουργία του είναι ιδιαίτερα επιβοηθητικός για να μειωθούν οι αποκλήσεις μέσω του ενιαίου χειριδίου Συγγνώμη αν ε, Παρακαλώ ολοκληρώστε γιατί δεν έχω χρόνο. Ίσως απαντώντας σε μια περτέρα ερώτηση. Η Κέιτ Σουίνμπερν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Φάρκας. Νομίζω ότι όλοι κατανοούμε ότι προσπαθούμε να καταρτήσουμε κανόνες συνεννόησης μεταξύ κοινοβουλίου, διαπραγματευτικής κοινοβουλίου και των δικών σα αρμοδίων, καθώ και των υπόλοιπων αποπτικών αρχών και βεβαίω έχουν βελτιωθεί τρόποι συνεργασία μα ως τώρα. Απλώς με ενδιαφέρει τι βήματα θα κάνετε, τι θα γίνει όταν το κείμενο του επίπεδου 1 έχει περατωθεί. Η ομάδα σας καταλαβαίνει πλήρως τις πολιτικές προθέσεις των διαπραγματευτών ή θα βασιστεί στην νομική ερμηνεία της εγγλικής εκδοχής του κειμένου. Έπειτα, πώς σκοπεύεται η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής μας να γνωρίζουν τις δράσεις που θα καταρτήσετε για την ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών και ερωταπαντήσεων και έπειτα πώς σκοπεύετε να ε, παρουσιάσετε τα απορίσματα του παρακολούθησης για την σύγκληση ως προς την υλοποίηση κυρίως. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις για την ερμηνεία του κειμένου του επίπεδου 1 και τις πολιτικές προθέσεις των συνομοθετών θα πρέπει να ε, επαφιόμεθα στις συμβουλές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ατύπω δεν είμαστε, επισήμω μάλλον δεν είμαστε μέρο του τριμερού διαλόγου, οπότε μέχρι να ολοκληρωθεί το κείμενο επίπεδο 1 βασιζόμαστε στην Επιτροπή. Έπειτα για την ε, αφοσίωση του Κοινοβουλίου και το τι θα γίνει με το θέμα των ερωταπαντήσεων, όντω ανέκαθεν ήμασταν έτοιμοι για να συζητήσουμε, να συνεχθούμε με το Κοινοβούλιο για τα θέματα προτεραιότητε στην κατάρτιση και την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και κατά διαδικασία ε, σύνταξης των κειμένων ή την ε, φάση των διαβουλεύσεων ή τη φάση της, του ελέγχου των κειμένων. Στις ερωταπαντήσεις έχουν δοθεί ε, αρκετά στοιχεία. Αλλά στην όλη αυτή διαδικασία και όταν τα θέματα που είχαν να κάνουν με τα θέματα ερμηνείας στο επίπεδο 1 η Επιτροπή πάντοτε είχε συμμετοχή ιδίω τα θέματα συντονισμού επίπεδου 1 και του επίπεδου 2. Και σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να ε, έχουμε κάπως ευρύτερες ερωταπαντήσεις για την σύγκληση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημοσιεύσουμε μια σειρά από εκθέσεις όπως τις εκθέσεις ομοτήμων ή την θεματική ανάλυση των προσπαθειών ε, σύγκλησης και στον ε, κρατικό τομέα αυτό είναι μια σαφής ένδειξη για το πώς η πρόοδος έχει καταβληθεί σχετικά. Κάνουμε και πολλή δουλειά που δεν δημοσιοποιείται για τις συναντήσεις διαμεσολάβησης σε επίπεδο ομαδικό, κάτι που δεν θα μπορούσαμε να δημοσιεύσουμε. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκίγκολντ. Με συγχωρείτε, δεν ήξερα ότι ήταν ε, άλλο εδώ στη θέση του. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη, Πρόεδρε. Κύριε Φάρκα, καλημέρα σα. Πρώτα απ' όλα τι απόψει σα για τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν αποδοθεί στι Ευρωπαϊκέ εποπτικέ αρχέ. Θα ήταν ε, καλό να έχουμε κάποιο ποσό για να καλύπτουμε ένα μέρο του προπολογισμού του. Κάποιε αμοιβέ. Και έπειτα για την μεθοδολογία εργασία των εποπτικών αρχών. Πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ εθνικών εποπτών και ημών και υπάρχει διαχωρισμό μεταξύ μελών της Ευρωζώνης και μη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Για να απαντήσω στην πρώτη, νομίζω ότι να προβλέψουμε αμοιβέ για τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών είναι κάτι που το σκεφτόμαστε αυτόν το καιρό και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει ίσως να ανακουφίσει κάποια από τα βάρη χρηματοδότησης τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Ίσως λοιπόν και εν μέρη να ήταν μια λύση. Το δεύτερο σημείο. Η συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών και των εθνικών αρχών και ενδεχόμενος ε, διαχωρισμός των εντός και εκτός ευρωζώνης. Η δομή μας βασίζεται στην εκπροσώπηση των εθνικών αρμοδίων αρχών. Μια αρχή λοιπόν της EBA από κυβερνητική και μόνο μορφή είναι απόφαση των μελών του Συμβουλίου που έχουμε μέλη των εθνικών αρμοδίων αρχών. Εξορισμού λοιπόν ο συντονισμός υπάρχει. Και επίση να θυμίσω ότι είπε και ο Ανδρέα Αρία για το θέμα αυτό. Υπάρχει κάποιε φορέ διαχωρισμό μεταξύ των διαφόρων εθνικών συμφερόντων και τη ευρωπαϊκή άποψη, την οποία μπορεί να εκπροσωπούμε εμεί οι απόψει του προσωπικού μα και των συνεργατών μα, όμω αυτέ οι διαφωνίε τις περισσότερε φορέ μπορούν να γεφυρωθούν αρκετά απλά. Ως προ τι διαφορές για του όσου είναι εντό και εκτό ευρωζώνη, να πω ότι ως τώρα η διαφορά αυτή τουλάχιστον στο τραπεζικό εγχειρίδιο κανόνων, στους τραπεζικούς κανόνες, δεν είναι τόσο έντονη, τόσο ορατή όσο κάποιοι έχουν περιγράψει. Έτσι όπως το έχουν δηλαδή περιγράψει τα μέσα ενημέρωσης ή ε, κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με όλους, ασχέτως αν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Ευχαριστούμε κύριο Γκίγκολτ. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα στο τομέα των αρμοδιοτήτων σας συγκεκριμένα να μου πείτε εάν η ΕΤΑ έχοντας κάποια εμπειρία από τη, διάδοση, από τη διάθεση στον κλάδο εγγράφων θα ήταν ε, διατεθειμένη να προχωρήσει σε ένα καθεστώς μεγαλύτερη διαφάνεια στη σχέση της με τον κλάδο, γιατί βλέπουμε ότι μπορεί η ηγεσία να το υποστηρίζει αυτό, αλλά το προσωπικό έχει, πέραν των διαβουλεύσεων, επαφές σε άτυπο επίπεδο, σε άτυπη βάση με τον κλάδο. Και γι' αυτό ερωτώ εάν η ΕΤΑ είναι δετεθειμένη να προχωρήσει σε μια ευρεία κλίμακο ε, διαδικασία διαφάνεια διαδικασίας διαφάνειας στη σχέση με τον κλάδο. Απάντηση. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε σαφώς ε, δεσμευθεί για απόλυτη διαφάνεια στις επαφές μας με τον κλάδο. Αυτό πράττουμε διαρκώς. Βεβαίω με τις διαβουλεύσεις έχουμε επαφές, αλλά αυτές είναι δημόσιες ε, εκδηλώσεις. Και έχουμε στήσει από το προσωπικό μας να καταγράφει οποιαδήποτε επικοινωνία με τον κλάδο. Και αν υπάρχει λόγος να διερευνήσουμε περαιτέρω κάποιες επαφές, το πράττουμε. Ναι, αλλά ερωτήσεις μπορεί να ε, διατυπώσει κανείς μόνο αν ξέρει ότι έγινε κάποια επαφή ή μια συνάντηση. Πώς ξέρετε εσείς ότι κάποιος από το προσωπικό σας είχε επαφές και συναντήσεις με εμπλεκόμενους προσώπους του κλάδου. Ε, αυτό προσπαθούμε να καταγράφουμε. Να κρατάμε ένα μητρό. Και αν δημοσιοποιηθεί τότε καλούμε τον εν λόγω υπάλληλο να απαντήσει αν ευσταθούν όλα αυτά που καταγράφονται ως πληροφορίες. Ευχαριστώ. Δεν μόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Κύριε Φάλκα, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας ένωσης για την αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων για τις τράπεζες, ε, βλέπουμε το έργο της ΕΤΑ. Φυσικά εμείς ως πατριώτες υποστηρίζουμε το έργο των εθνικών υποπτικών ε, αρχών, αλλά δεδομένη της ε, σοβαρότητας οικονομικής κατάστασης θεωρούμε ότι πρέπει να υποστηρίζετε και το δικό σας έργο. Ωστόσο, οι αμοιβέ των τραπεζιτών δεν τηρούν τους ισχύοντες κανόνες και ο, της εκπλήξεως αυτοί οι τραπεζίτες ε, είναι οι κατεστημένοι επιτοπλίστων στο Λονδίνο. Χρόνια τώρα συνεχίζεται η παρανομία αυτή και πρέπει να τεθεί τέρμα. Και ενώ η ΕΚΤ διαθέτει δισεκατομμύρια ευρώ για να διασώζει τις τραπεζικές, ε, ε, τα τραπεζικά ιδρύματα εδώ και χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι έχουν απίστευτα υψηλές αποδοχές και αποζημιώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να Συνεχίζει την παρανομία εδώ και τόσο καιρό και να είναι εγκατεστημένα στη ΣΥΤΗ τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Απάντηση. Ε, θα μου επαναλάβετε σα παρακαλώ το τέλος της ερώτησής σα γιατί δεν ήταν τόσο σαφής. Ναι, πώς γίνεται η πλειονότητα των τραπεζών αυτών που παρανομούν να είναι τράπεζες του ΣΥΤΗ. Απάντηση. Καταρχάς, νομίζω ότι έθιξα το έργο της ΕΤΑ ως προς τις αμοιβέ και αποδοχές και τις εκθέσεις μας. Δεύτερον, για τα σχόλιά σας. Όντως πιστεύω ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προβεί σε σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση του λεγόμενου ηθικού κινδύνου ε, δηλαδή της ε, ανάγκης για διάσωση από, την, ε, από τον νομοθέτη της, των τραπεζών που στηρίζονται σε τέτοιες συνθήκες. Και βέβαια το, όλο σύστημα εκαθάρισης, εξυγένσης καλύτερα, έχει να κάνει με τον ηθικό κίνδυνο. Τώρα, το ποιοι είναι αυτοί οι φορείς οι οποίοι έχουν έδρα και πού, όλοι ξέρουμε ότι το Λονδίνο και το City συγκεκριμένα είναι κύριο χρηματοπιστωτικό κέντρο. Οι τράπεζε οι οποίε υπάγονται στι ρυθμίσει ε, για τι αμοιβέ, κατευθυντήριε γραμμέ για τι αμοιβέ και τι αποδοχέ, ε, οφείλουν να τηρούν του ίδιου κανόνε ανεξαρτήτω τη έδρα του. Εάν λοιπόν δούμε ότι ξεφεύγουν από τον κανονισμό, Εάν δεν είναι στο πεδίο δράσεω τη ΕΤΑ ή συγκεκριμένου κανονισμού, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ. Έτσι καταλήγει και αυτή η συγκεκριμενου κανονισμου δυστυχω δεν μπορουμε να Ευχαριστούμε πολύ. Welcome Καλώς ήρθατε κυρία Βερίνα ε, Ρος που είστε εκτελεστική διευθύντρια του ΕΣΜΑ και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ανυπομονώ να συζητήσουμε για τη μελλοντική πορεία της ΕΣΜΑ και να εξηγήσω, γιατί θα ήθελα να είμαι εκτελεστική διευθυντήρια και σε αυτές τις στιγματικές ε, μέρες λειτουργίας της ΕΣΜΑ. Κοιτάζοντας προς το παρελθόν, θεωρώ ότι συνολικά η ΕΣΜΑ έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με τους βασικούς της στόχους και την ίδρυσή της το 2011. Όπως είπε προηγουμένως ο Στίβεν, αυτή η θετική αποτίμηση έχει επιβεβαιωθεί από εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης από το 2014. Το ίδιο και με την έκθεση τη πρωτοβουλίας που συντάξετε εσείς. Ε, είχαμε το ενιαίο χειρίδιο κανόνων, το εποπτικό σύστημα για τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους, την ανάλυση του κινδύνου και τα σημαντικά βήματα για την εποπτική σύγκληση. Όλοι απαιτητικοί στόχοι. Αυτά μας επέτρεψαν να έχουμε καλύτερη προστασία των επενδυτών, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εύρωστε αγορέ, δηλαδή του βασικού μα στόχου. Έχουμε μεγαλώσει και καλύτερα ε, λειτουργούμε ω μια ε, εύρυθμη αρχή που λειτουργεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην καθημερινότητα της ΕΣΜΑ έχουμε από την αρχική ίδρυση και πρόσληψη της ε, ομάδας των συνεργατών την διαχείριση του προπολογισμού της ΕΣΜΑ, τους πόρους που αφορούν τον προπολογισμό, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εκτέλεση του προγράμματος δράσης μας και προσωπικά αυτά είναι και τα βασικά θέματα που με απασχολούν. Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία ήταν ε, γεμάτα ε, θετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια και προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες ιδίως με την περίπτωση της ΕΣΜΑ. Το να εργαζόμαστε λοιπόν για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και για την Ευρώπη ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Βεβαίως η πορεία για το μέλλον δεν θα είναι απλή. Έχουμε διαγράψει στου στρατηγικού προσανατολισμού της ΕΣΜΑ και το σχετικό έγγραφο τη θεώρησή μας για το μέλλον. Έχει δημοσιευτεί ήδη στις αρχές τη χρονιά. Έχουμε το εγχειρίδιο, το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων που ευτυχώ ολοκληρώνεται και περνάμε τώρα στο κεφάλαιο υλοποίηση. Έχουμε συμβάλει ιδιαίτερω στα ρυθμιστικά θεμέλια επί των οποίων θα οικοδομήσουμε για να έχουμε μία ε, ενιαία κεφαλαία αγορά στην Ευρώπη με οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση όπω ε, οι ανάγκε τη Ευρώπη ορίζουν και μετά από αυτήν την ένωση και το πρόγραμμα δράσης που έχουν εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά ως έσμα μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Όμω, πολύ σύντομα να μιλήσω για τι προκλήσει υλοποίηση σε τρει συγκεκριμένου τομεί. Πρώτα απ' όλα, η υλοποίηση. Θα χρειαστεί να έχουμε την οικοδόμηση και εύρυθμη λειτουργία συστημάτων πληροφορική για να συλλέγουμε δεδομένα και να δημοσιεύουμε τι απαραίτητε πληροφορίε που θα επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι αγορέ τη να λειτουργήσουν επιτυχώ. Η αρμόδιες ελληνικέ αρχέ από 27 χώρε. έχουν συμφωνήσει να εκχωρήσουν την οικοδόμηση και λειτουργία κάποιων ε, συστημάτων πληροφορική σε σχέση με την οδηγία MIFID 2 στην ΕΣΜΑ. Η αρχή γίνεται λοιπόν ουσιαστική σημασία στην ε, υποδομή, τη διάρθρωση των συστημάτων για τις ευρωπαϊκές πυθαλαγορέ και την ίδια την αγορά και τη λειτουργία τη θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τις δυνατότητές μας πληροφορική με ένα ε, επιτυχημένο πρόγραμμα του παρελθόντος θα πρέπει να επαναληφθεί βεβαίω για να είμαστε επίκαιροι και να δίνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές. Η υλοποίηση επίσης θα, ε, θα μας ε, απαιτήσει να ευθυγραμμίσουμε τα αποτελέσματα και τις πρακτικές των εποπτών. Με το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αναπομένασεις ε, παρεκκλήσεις για να έχουμε τη σωστή διαμεσολάβηση και να μην υπάρχει πλέον κατακαιρματισμός της αγοράς. Έχουμε ένα λεπτομερέστατο πρόγραμμα εργασίας για την εποπτική σύγκληση ε, για το 2016 το οποίο θα συμπληρώσει το ε, γενικότερο πρόγραμμα εργασίας και το πολυετές που ήδη έχουν δημοσιευτεί για την εποπτεία από από κάποιους μήνες. Θα πρέπει να έχουμε τι απαραίτητες δυνατότητες και να αξιοποιήσουμε την μέχρι τώρα εμπειρία μας στην μετατόπιση της δουλειάς μας από την εποπτεία, στην σύγκληση αυτό θα σημαίνει νέα επικέντρωση των προτεραιότητων μας, αλλά για κάποιες προκλήσεις ως προς τους ανθρώπινους πόρους στην κατάρτιση και την εσωτερική κινητικότητα. Επίσης θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται αυτή τη στιγμή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταλαβαίνουμε, αναλύουμε και αναχαιτίζουμε καλύτερα τους κινδύνους που μπορεί να εμποδίσουν την επιτεύξη των στόχων της ΕΣΜΑ. Η καλύτερη χρήση των δεδομένων σημαίνει η συλλογική προσπάθεια από την ΕΣΜΑ και άλλους φορείς της ΕΕ, Ένωσης όπως η Μικτή Επιτροπή των Εποπτικών Αρχών, η ΕΣΑΡΜΠΗ και ούτω καθεξής, καθώς και στενή συνεργασία με τι ε, εθνικές αρχέ. Για να μπορέσει η ΕΣΜΑ να διαδραματίσει αυτό το ρόλο, ε, αλλά και να αντιμετωπίσει και τις επόμενες προκλήσεις του μέλλοντος, θα πρέπει να έχουμε ένα σταθερό και ισχυρό οργανισμό. Ο ρόλος μου ως εκτελεστική διευθυντής θα είναι να συνεχίσω να επικεντρωνομαι στην πρόσληψη, την ε, εκπαίδευση και την διατήρηση των εξαιρετικών συνεργατών, με σωστέ προτεραιότητε για το πρόγραμμα εργασία τη ΕΣΜΑ, υψηλή ποιότητα και, επίκαιρη, και έγκαιρη επίτευξη αποτελεσμάτων. Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε την στήριξη της Επιτροπής ΕΚΟΝ και των μελών της, αλλά θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον όπου οι προπολογισμοί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Εθνική θα περιορίζονται, θα συμπιέζονται διαρκώς. Γι' αυτό θα συνεχίσω την διαχείριση της ΕΣΜΑ με τρόπο διαφανή, δίνοντας προτεραιότητα τα αποτελέσματα που επιθυμούμε να πετύχουμε με το πρόγραμμα εργασία μα. Είμαι ευγνώμων και ικανοποιημένη που το ε, Συμβούλιο Εποπτών τη ΕΣΜΑ ε, προέβλεψε την ε, παράταση τη θητεία μου για άλλα πέντε χρόνια. Δεν θα είναι ένα εύκολο διάστημα, αλλά μετά τι προκλήσει των προηγούμενων 4,5 ετών, ευχαρίστω να αντιμετωπίσω τι προκλήσει και ευκαιρίε του ερχόμενου διαστήματο με τον Στίβεν και του συναδέλφου μου. Ελπίζω να πετύχουμε ω ΕΣΜΑ. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Παύλο Σάλβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Ρος για την παρουσία σας. Πρώτα απ' όλα να είμαι λίγο επικριτικός για το MIFID, για την οδηγία MIFID. Ξέρετε ότι είναι βασική σημασία για το σώμα μας. Και το Κοινοβούλιο δεν είναι πολύ ικανοποιημένο με την πρόταση να αναβληθεί η ε, εφαρμογή, του, εφαρμογή της για άλλο ένα χρόνο, γιατί έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια από τότε που εγκρίθηκε το κείμενο από τους συνομοθέτες. Ε, Αν είχε λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η ΕΣΜΑ, δεν θα αρκούσαν τα τρία χρόνια. Και τι διδάγματα εξάγεται από αυτή την καθυστέρηση. Τι θα επιχειρήσετε να αποφύγετε στο μέλλον, εάν βεβαίως επικυρωθείτε. Επίσης, τι φταίει για αυτή την καθυστέρηση καθυστερήσεις και στην ΕΣΜΑ και στην Επιτροπή υποθέτω. Θα ήθελα όμως τη γνώμη σας. Γιατί το Κοινοβούλιο εγκαίρως επετέλεσε το καθήκον του. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για την καθυστέρηση. Κάτι άλλο για την Ένωση των Κεφαλαίων που αναφέρατε εδώ στην εισαγωγική συνομιλία. Θα γνωρίζετε την πρόταση της Επιτροπής για την τιτλοποίηση η οποία είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη από το σώμα μας. Η Επιτροπή μας τις επόμενες εβδομάδες θα συζητήσει τροπολογίες από αυτής της προτάσεις. και ξέρετε ότι μία από τις ανησυχίες μας αφορά την ε, χρηματοδότηση των μικρομεσιών. Θεωρείτε ότι θα επαρκέσει η πρόταση της Επιτροπής για αυτή τη χρηματοδότηση. Γιατί εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Όχι παρακαλώ, παρακαλώ πρόεδρο. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. όχι. Ε, παρακαλώ, δύο ερωτήσει. Αρκούν. Απάντηση για την καθυστέρηση της ΜΥΦΙΔ. Κοιτάξτε, εργαστήκαμε πολύ αποδοτικά και ταχαίως για να ολοκληρώσουμε το σύνολο των μέτρων, το τεράστιο σύνολο μέτρων επίπεδου 2 και το καλοκαίρι, αποφασίσαμε να καθυστερήσουμε για ένα τρίμηνο την υποβολή των προτάσεων για να γίνει η αναγκαία νομική αποτίμηση και για να είναι και πιο ομαλή μετά η διαδικασία έγκρισης. Είναι απόλυτα σαφέ, Θεωρώ. Και το είπαμε και στην Επιτροπή ότι υπάρχουν θέματα για την ανάπτυξη της πληροφορικής και των συστημάτων και όλα αυτά παίρνουν τον χρόνο τους ούτως ώστε η ΜΥΦΙ 2 να λειτουργήσει αποτελεσματικά από την πρώτη μέρα που θα εφαρμοστεί που θα ισχύσει. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό προτείνουμε μια ενδεχόμενη καθυστέρηση, αλλά με πολύ σαφείς στόχους για να σκεφτεί η Κομισιόν τις προτάσεις πριν τις υποβάλει στους συνομοθέτες, γιατί εσείς θα πρέπει να αποφανθείτε από αυτόν. Εμείς λέμε ότι η ανάπτυξη της πληροφορικής θα είναι πολύ δύσκολη σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ολοκλήρωση του ιδιαίτερα τεχνικού επίπεδου των προδιαγραφών και της τεχνικής φύσης για το δεύτερο θέμα. Οι προτάσεις τυπλοποίησης θα βοηθήσουν τη χρηματοδότηση πιστεύω ενδεχομένως των μικρομεσαίων αλλά δεν επαρκούν από μόνες τους αυτές τις προτάσεις. Νομίζω ότι η ενιαία κεφαλαία έχει και άλλες προτάσεις για να στηρίξει τις μικρομεσαίες. Ελίζα Φερέρα. Ευχαριστώ, δεν έχω χρόνο για να σας επενέσω για αυτά που έχετε κάνει περισσότερο. Για την ένωση των κεφαλαιοαγορών είναι πολύ χαμηλά τα επιτόκια, είναι η κίνδυνοι. Θεωρείτε ότι το νέο εγχειρίδιο είναι επαρκές για να αντιμετωπίσει τους νέους κινδύνους. Δεύτερον, πώς βλέπετε το ρόλο σας ως ε, εποπτικού φορέα στα πλαίσια των νέων προκλήσεων που θα δημιουργήσει η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Θεωρείτε ότι χρειάζεται πλέον αρμοδιότητες ή αρκούν. Απάντηση. Ευχαριστώ για το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Οπωσδήποτε σημαίνει ότι υπάρχουν νέοι κίνδυνοι. Όλοι ψάχνουν δηλαδή να βρουν κερδοφορία κάπου και αυτό δημιουργεί κάποιους κινδύνους στην αγορά, τους οποίους επιτηρούμε πολύ προσεκτικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα ότι δεν επαρκεί το ενιαίο εγχειρίδιο. Κάποιοι κανόνες ακόμη βέβαια σταδιακά διαμορφώνονται. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα περάσουν στο εγχειρίδιο. Αλλά κυρίως πρέπει να επιβλέπουμε πού μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι και να βρούμε τις σωστές αντιδράσεις. Για τη δεύτερη ερώτηση της εποπτείας. Όπως ήδη είπα, το κύριο για μας είναι να προωθήσουμε σε όλη την Ένωση την ε, σύγκληση των συστημάτων εποπτείας για να έχουμε την ε, ενιαία την Ένωση και Κεφάλαια Αγορών χρειάζεται σύγκληση και της εποπτείας τους. Αυτό θα μας απασχολεί στα τα επόμενα χρόνια. Θα δούμε αν γι' αυτό χρειάζονται περαιτέρω θεμελιώδεις αλλαγές επειδή νομίζουμε ότι πολλά από τα μέσα που χρειαζόμαστε τα έχουμε. Και θα δούμε και του επόμενου μήνε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε κυρία Σουίμπερν. Ευχαριστώ και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτική. Ήδη έχω συγχαρεί την ομάδα. Πάντως πρέπει να γνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην νομοθεσία διότι υπήρξαν παρανοήσεις για τις πολιτικές προθέσεις των διαπραγματευτών. Και όχι μόνο για την ερμηνεία των ε, νομοτεχνικών για την τελική μορφή των κειμένων. Πώς πιστεύετε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, ώστε η ομάδα έσμα, της ΕΣΜΑ να καταλαβαίνει πλήρως το ότι υπονοούν αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να πρώτο αρχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά για τα ATS, δηλαδή τα τεχνικά πρότυπα ρύθμισης στην πράξη. Μήπως πρέπει να γίνεται κάποιο είδους απενημέρωση προηγουμένως και επίσης για τις δυνατότητες πληροφορικής που έχετε. Είπατε ότι τώρα θα έχετε τεράστιο όγκο δεδομένων και θα πρέπει να τα αναλύετε, να τα επεξεργάζεστε. Έχετε τα απαραίτητα εργαλεία, θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό με το σύστημα ε, πληροφορικής ή θα πιάσουν σκόνη αυτά τα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα. Να πω ότι είναι σημαντικό για μας να κατανοήσουμε τις πολιτικές προθέσεις κάποιων από τις τελικές συμβιβαστικές προτάσεις, ιδίως στη δικασία επίπεδου 1, διότι προφανώς για μας προτεύει να μπορούμε να εργαστούμε στο επίπεδο 1 για να υλοποιήσουμε ικανοποιητικά τα μέτρα του επίπεδου 2. Και με εσά λοιπόν και με το Συμβούλιο ο στόχος ήταν να κατανοήσουμε. Να κατανοήσουμε αν και αυτή τη στιγμή ε, επαφιόμαστε περισσότερο στην Επιτροπή που είναι ο συνομιλητής μας στην διαδικασία καθ' τη διάρκεια αυτής. Όμως θα ήταν ε, καλό να ενημερωνόμαστε και για τις συζητήσεις στο επίπεδο 1. Θα μας εξυπηρετούσε πολύ για να καταλάβουμε καλύτερα. Ως προς τα θέματα υπολογής των πληροφορικής υπάρχουν εδώ δύο βασικές προκλήσεις. Η εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζεται για να χτιστεί το σύστημα και να λειτουργήσει όρθος και αποτελεσματικός ε, και αυτό για να μπορέσει η οδηγία να εφαρμόζεται αμέσως ε, αποτελεσματικά. Μετά το άλλο θέμα είναι οι δυνατότητες επεξεργασίας και ανάλυσης που έχουμε εσωτερικώς και πώς μπορούν τα δεδομένα που θα αναλυθούν να αξιοποιηθούν. Βεβαίως υπάρχει πίεση εδώ, δεν θα το κρύψω. Έχουμε πολύ καλούς εμπειρογνώμονες που είναι σε θέση να τα κάνουν όλα αυτά, όμως θα να δώσουμε προτεραιότητα στη δραστηριότητα αυτή με μεγάλη προσοχή και σύνεση. Δεν έχουμε τόσους πολλούς πόρους όσο θα θέλαμε ιδανικώς για να κάνουμε όλη τη σωστή ανάλυση όλου του τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε στενά με τις εθνικές αρχές, γιατί εκείνοι θα συγκεντρώνουν σε εθνικό επίπεδο κάποια δεδομένα ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ. Κύριε Χάρκιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Και καλημέρα σας. Σύντομα. Συμφωνείτε με τον κύριο Φάρκας σε σχέση με τα οικονομικά μέσα που έχουν στη θέση τους οι εποπτικές αρχές. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιβληθούν τέλη για να καλύπτονται κάποιες από τις ανάγκες σας και ο προπολογισμό σας. Δεύτερον, πώς βλέπετε το ρόλο σας ε, στην παγκόσμια διακυβέρνηση και το ρόλο της Επιτροπής σε σχέση με το δικό σας ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, για τη χρηματοδότηση και την επιβολή τέλους. Ε, σε ένα βαθμό η ΕΣΜΑ χρηματοδοτείται από τέλη που συλλέγουμε από τις εταιρείε αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου. Ένα τρίτο λοιπόν της χρηματοδότησης μας προέρχεται από αυτές τις πηγές. Και πιστεύουμε ότι υπάρχει όντως ε, περιθώριο να εξετάσουμε την περαιτέρω επέκταση της χρηματοδότησης αποτέλει, όχι μόνο για την ΕΣΜΑ, αλλά για όλες τις υποπτικές αρχές, ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους. Επίσης, για να πέρασω στη δεύτερη σας ερώτηση για την ΑΙΟΣΚΟ, είμαστε παρατηρητές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΙΟΣΚΟ και προφανώς με συγκεκριμένους όρους και στοχευμένα προσπαθούμε να συμβάλλουμε στο έργο της ΑΙΟΣΚΟ στο βαθμό που αφορά το ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Δεν μπορούμε να καλύψουμε κάθε θέμα, αλλά όπου χρειάζεται, όπου είναι πιο σκόπιμο, το πράττουμε. Και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Φυσικά είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και με την Επιτροπή εν γέννη ως προς τη δράση μας σε διεθνείς ε, χώρους συναντήσεων και συνομιλιών. Είναι προφανές ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει με μία φωνή στη εθνική κοινότητα. Ευχαριστώ, κύριο Κίκολτ. Πολύ σύντομα και καλημέρα σας. Αλλά η θετική απάντηση της ΕΤΑ για τις ε, συνέπειες της άνησης προσφοράς πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναντι εκείνων που παρέχονται σε εκπροσώπους του κλάδου. Με εμπνέει να υποβάλω αντίστοιχα ερώτημα και στην ΕΣΜΑ. Έχετε κάποια απάντηση για να εξασφαλίσετε διαφάνεια αντί των λόμπι και για το προσωπικό σας εκτός των διαβουλεύσεων με έναν κατάλογο ενδεχομένω που θα δημοσιοποιείτε για το ποια είναι τα λόμπι με τα οποία έχετε επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση και ίσως και μια πρώτη αντίδραση για το γεγονός ότι για το γεγονό που έχουμε συστήσει και στο παρελθόν, ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση ε, εναντί αυτών. Ναι, νομίζω ότι ο κύριο Φάρκα απάντησε στο ερώτημα της άνησης πρόσβασης. Είναι πολύ ατυχές αυτό και βεβαίως πρέπει να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μα ώστε οι πληροφορίε που πρέπει να δημοσιοποιούνται να διατηθούνται στο κοινό και εκείνες που δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται να παραμένουν απόρριτες. Ε, όπως ξέρετε ήδη έχουμε δημοσιεύσει τις επαφές μας με τους εμπλεκόμενους παράγοντες και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Ε, με πόσο σκόπιμο από την ε, σκοπιά της αναλογικότητας είναι να δημοσιεύεται κάθε μία επικοινωνία και επαφή με εκπροσώπους, όχι μόνο του χρηματοπιστωτικού κλάδου, γιατί αν το κάνουμε πρέπει να το κάνουμε για κάθε εμπλεκόμενο φορέα και σε τελευταία ανάλυση το προσωπικό μας δεν έχει δουλειά ε, δημοσίων σχέσεων, έχει άλλο ρόλο να επιτελέσει. Από την άλλη, αν θεωρεί ευρύτερα το Κοινοβούλιο ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, μπορούμε να το ξανασυστήσουμε. Από την Επιτροπή δεν βλέπουμε να ισχύει κάτι αυτή τη στιγμή για το προσωπικό της αλλά αν θέλει το κοινοβούλιο να αλλάξει η πολιτική, πολύ ευχαριστώ να το συστήσουμε. Λοιπόν, τελευταία η Μπάρμπαρα Κάπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Ρώση, για την παρουσίασή σας. Να αναφερθώ στο MIFID, πολύ συγκεκριμένα και ειδικά. Τροπολογία των ε, ρυθμίσεων για τις παράπλευρες δραστηριότητε. Αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τις εταιρείες που ασχολούνται με τις πρώτες ύλες και ιδιαίτερα για τον τομέα της ενέργειας. Ορισμένοι εξαιρέθηκαν από το MIFID. Αυτή η νέα ρύθμιση όμως σημαίνει μεγάλες υποχρεώσεις για υψηλότερο κεφάλαιο και την τήρηση ορισμένων ε, ε, μέτρων για την υποβολή ισολογισμών. Γιατί η ΕΣΜΑ ε, δεν υποστηρίζει τον κανονισμό που αυτή τη στιγμή δεν, ε, δεν, δεν στηρίζει τον κανονισμό που δεν επιτρέπει καμία εξαίρεση. Και τι λέει η ΕΣΜΑ, για το ποσοστό που αναφέρεται για τις παράπλευρες δραστηριότητε. Ευχαριστώ πολύ. Εργαστήκαμε πολύ για αυτό το θέμα της MIFID όπως και για άλλα τμήματα. Η δραστηριότητα η παράπλευρη δραστηριότητα και το τεστ για, την, για το καθορισμό της παράπλευρης δραστηριότητας ήταν πολύ δύσκολος τεχνικά για την εργασία μας ε, για το επίπεδο 2 της MIFID. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο για να μετρήσουμε ποιοι είναι πραγματικά σημαντικοί συνολικά για την αγορά ή και εάν και σε κατά πόσο η δραστηριότητα αυτή παράπλευρη είναι σημαντικό τμήμα της συνολικής τους δραστηριότητας και προσπαθούμε ο ορισμός να διαμορφωθεί έτσι ούτως ώστε να αφορά μόνο εκείνους που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά που έχουν σημαντικές επιπτώσεις ε, σε μια αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος μια συγκεκριμένης πρώτης ύλη. Θα δούμε τώρα τι επιπτώσεις θα έχει. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχει πολλές επιπτώσεις σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Θεωρούμε όμως ότι είναι αρκετά θεμητός ο ανταγωνισμός για τις επιχειρήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που είναι ενεργοί και σε αυτές τις αγορές πρώτων υλών και για μερικές βασικές επιχειρήσεις που είναι οι κυριότερες σε αυτό το τομέα και σε αυτές τις αγορές κάποιων ε, πρώτων υλών και που δεν υπάγονται στο ίδιο κανονιστικό πλαίσιο. Προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε μπορεί να καταλήξει και αυτή η τελευταία ακρόαση που ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Σας ευχαριστώ και πάλι και όλους τους συναδέλφου σας. Ευχαριστώ και τους άλλους Προέδρους για αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε την κρίση μας. Η ψηφοφορία για την ολοκλήρωση της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αναβλήθηκε για την 1η Δεκεμβρίου, οπότε μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου και φυσικά θα συνεδριάσουν ε, οι συντονιστές για να αποτιμήσουν ε, τις ακροάσεις μας που θα, και θα αποτελέσει αυτή η συζήτηση τη βάση των συστάσεων που θα ψηφίσουμε την 1η Δεκεμβρίου στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια του Στρασβούργου το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τους τρεις ε, προέδρους και τους δύο εκτελεστικούς διευθυντές. Λίγη συνεδρίαση.